Θα αρχίσουμε τις εργασίες μας με το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης, το 17, να καλωσορίσουμε τους δύο εκπροσώπους της Βουλγαρικής Προεδρίας. Πρόκειται την κυρία Σάσεβα που ε, είναι Υπουργός Δικαιοσύνης και τον κύριο Πολουμπανόφ που είναι Υπουργός Πολιτισμού που θα μας μιλήσουν για τα βασικά σημεία του προγράμματος που τους απασχολεί και θα μας μιλήσουν για την ε, Βουλγαρική Προεδρία και τις προτεραιότητες της. Έχετε 20 με 25 λεπτά τα οποία μπορείτε να μοιραστείτε όπως θέλετε. Δηλαδή 15 λεπτά ε, καστός διότι στην Επιτροπή μας στη συνέχεια οι βουλευτές θα σας υποβάλουν ερωτήσεις. Έχετε το λόγο κύριε μου. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε μέλη του Ευρωκοινοβουλίου. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για αυτή την ε, δυνατότητα που μου δίνετε να ασχοληθώ με τα βασικά ζητήματα της ε, ατζέντα μας και τις βασικές προτεραιότητες στον τομέα της δικαιοσύνης. Οι θετικές εξελίξεις όλων των τομέων που άπτονται της δικαιοσύνης σχετίζονται με την συνεργασία με τη δική σας Επιτροπή. Με την ευκαιρία αυτή θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και, τους, και εσάς και τους συναδέλφους της Εστονικής Προεδρίας για την κοινή εργασία μας και πιστεύω ότι η Βουλγαρική Προεδρία μαζί με τα κράτη-μέλη ε, αυτής της ε, τριάδας προεδριών θα φτάσουν σε λειτουργικές λύσεις και επικοδομητικές. Εμείς αναλαμβάνουμε το πιδάλιο του Συμβουλίου τη στιγμή που οι μελλοντικές εξελίξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξαρτώνται από την ενότητα και αλληλεγγύη των κρατών μελών. Θα συνεργαστούμε για να προωθήσουμε μία ε, εύρωστη και ε, Ενωμένη Ευρώπη με βάση την ανταγωνιστικότητα και τη συνοχή. Η ευημερία και η ανάπτυξη θα πρέπει να αποτελέσουν βασικές μας αρχές. Τήρηση θεμελιωδών δικαιωμάτων και επικράτηση του κράτους δικαίου. Μία από τις βασικές προτεραιότητες για τη Βουλγαρική Προεδρία είναι ο νέος κανονισμός ε, ε, Βρυξέλλες 2α. Έχει μεγάλη σημασία για πληθώρα Ευρωπαίων πολιτών και αφορά ευαίσθητες πτυχές της καθημερινής του ζωής. Γονική ευθύνη, ε, απαγωγή παιδιών και ούτω καθεξής. Πρόκειται για αναδιατύπωση του υπάρχοντος κανονισμού Βρυξέλλες 2α που αποτελεί ένα από τα βασικά μέσα στον τομέα του οικογενειακού δικαίου. Άρα στόχος μας είναι να θέσουμε σε εφαρμογή αυτό το κανονιστικό πλαίσιο. Δέκα χρόνια μετά από τη θέση σε εφαρμογή αυτού του κανονισμού έγινε μια αξιολόγηση της εφαρμογής του και τα αποτελέσματα αυτής της αξιολόγησης δείχνουν ότι παρά τα θετικά αποτελέσματα, δυστυχώς ε, υπάρχουν σοβαρά προσκόμματα. Γι' αυτό είναι αναγκαίο να τροποποιήσουμε τον κανονισμό, έτσι ώστε να βελτιώσουμε το νομικό πλαίσιο και να μπορέσουν οι πολίτες να ε, υποστηρίξουν τα δικαιώματά τους στον τομέα του οικογενειακού δικαίου. Επίσης, χρειάστηκε να λάβουμε υπόψη τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου από το 2016 υπάρχουν αποφάσεις, 20 στον αριθμό που άπτονται αυτό το τομέα του οικογενειακού δικαίου. Και αυτό καταδεικνύει την ανάγκη μιας αλλαγής και φυσικά δείχνει ότι υπάρχουν ακόμα θέματα προς επίλυση. Άρα η αναδιατύπωση του κανονισμού ε, Βρυξέλλες 2α αποτελεί μια ε, περίπλοκη διαδικασία, αλλά θεωρούμε πλέον ότι θα πρέπει να φτάσουμε σε μια συμφωνία στα θέματα ζωτικής σημασίας που άπτονται αυτού του ζητήματος. Η Βουλγαρική Προεδρία θα προσπαθήσει να συγκεράσει τις θέσεις των κρατών μελών. Θα προσπαθήσουμε να φτάσουμε σε βελτιστοποιημένες και δίκες λύσεις έτσι ώστε έχουμε ε, καλύτερες δικαστικές αποφάσεις έτσι ώστε να μπορούμε να ε, ακροαστούμε τα παιδιά εκεί που χρειάζεται ιδιαίτερα σε σχέση με τις διεθνείς απαγωγές παιδιών και να μπορέσουμε να συνεργαστούμε με τις αρχές των κρατών μελών. Πιστεύω ότι τα κράτη-μέλη θα μπορέσουν να φτάσουν σε μία συνένεση σε σχέση με το νέο προσχέδιο του τροποποιημένου κανονισμού και θα φτάσουμε σε μία εξισορροπημένη άποψη σε σχέση με την αμοιβαία εμπιστοσύνη προς συμφέρον του παιδιού. Επίσης, η Βουλγαρική Προεδρία θα υποστηρίξει τις μεταρρυθμίσεις για την προώθηση της οικονομικής και κοινωνικής σταθερότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και καταβάλουμε μεγάλες προσπάθειες για να βελτιώσουμε το νομικό πλαίσιο αφαιρεγγιότητας μέσα στα πλαίσια της αναδιάρθρωσης και διαδικαστιών δεύτερης ευκαιρίας. Το νομικό πλαίσιο επιτρέπει τους επιχειρηματίες να μπορέσουν να συνεχίσουν τις δραστηριότητες τους και έτσι θα μπορέσουν να συνεχίσουν με την εργασία τους έτσι ώστε να μην συρρυκνωθεί η εργασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα προσπαθήσουμε να φτάσουμε σε μία εξισορρόπηση του πλαισίου με κοινούς κανόνες για την αφαιρεγγιότητα και για τις διαδικασίες δεύτερης ευκαιρίας. Αυτή τη στιγμή συζητείται το όλο θέμα σε μια ομάδα εργασίας του Συμβουλίου και πιστεύουμε ότι κατά την Προεδρία μας θα φτάσουμε σε πρόοδο, ουσιαστική πρόοδο. Όσο αφορά το εταιρικό δίκαιο, θεωρούμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορέσει να εισαγάγει το νέο πακέτο μεταρρυθμίσεων και θα θέλαμε να ε, ασχοληθούμε το ταχύτερο δυνατόν με αυτό το πακέτο όταν τεθεί επιτάπητος. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η ανάπτυξη της ε, ενίας αγοράς για να λάβουμε υπόψη τα συστήματα των κρατών μελών που αποκλίνουν πολλές φορές. Επίσης, η ψηφιοποίηση του εταιρικού δικαίου θα μας απασχολήσει άμεσα. Θα λάβουμε υπόψη τη βούληση των κρατών μελών έτσι ώστε να έχουμε ένα, ένα στο νομικό πλαίσιο για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε την προσβασιμότητα σε αυτές τις ε, διαδικασίες έτσι ώστε να χρησιμοποιηθεί η ψηφιακή τεχνολογία για όλες τις ε, εμπορικές επιχειρήσεις. Σε σχέση με τις ΜΜΕ, που προσπαθούν να κινηθούν διασυνοριακά, θεωρήσαμε ότι πρέπει να εξυγχρονίσουμε τους κανόνες σε σχέση με τις διασυνοριακές συγχωνεύσεις για να εισαγάγουμε και νέους κανόνες σε σχέση με το ε, κατακαιρματισμό της αγοράς και την αλλαγή έδρας των εταιριών. Θα ήθελα να αναφέρω ότι μία από τις βασικές αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ελεύθερη κυκλοφορία, είναι ύψης της σημασίας για εμάς. Θα προσπαθήσουμε να εγγυηθούμε την προστασία των δικαιωμάτων όλων των εμπλεκομένων δηλαδή στο, όσον αφορά τους πολίτες, τις επιχειρήσεις, του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα και θα λάβουμε υπόψη και τους ε, κινδύνους των ε, πιστωτών, ε, επίσης και τον κίνδυνο φορολογικής απάτης και την ε, νομιμοποίηση παράνομου χρήματος. Στο τομέα του συμβατικού δικαίου θεωρώ ότι θα μπορέσουμε να φτάσουμε σε μία συμφωνία σε επίπεδο πρώτης ανάγνωσης σε σχέση με την παροχή ψηφιακού περιεχομένου. Όσον αφορά την πώληση αγαθών, θεωρώ ότι θα πρέπει να αρθούν τα προσκόμματα στο ηλεκτρονικό εμπόριο, ιδιαίτερα διασυνοριακά, και θα μπορέσουμε να βελτιώσουμε κατά αυτόν τον τρόπο το εταιρικό δίκαιο. Το συμβατικό δίκαιο, με συγχωρείτε. Αυτό που έχει σημασία είναι λοιπόν να δούμε την υποεκπροσώπηση των γυναικών σε επίπεδο λήψης αποφάσεων στα διοικητικά συμβούλια των επιχειρήσεων. Η Βουλγαρική Προεδρία θα προσέξει ιδιαίτερα αυτό το θέμα έτσι ώστε να μην υπάρξει αναστέλουσα μειοψηφία και να μπορέσουμε να προωθήσουμε αυτό το θέμα. Θεωρώ ότι όσον αφορά τις κοινωνικές ε, πολιτικές και την πολιτική απασχόλησης, θα πρέπει να συμφιλιώσουμε την ε, οικογενειακή και επαγγελματική ζωή, ιδιαίτερα αν λάβουμε υπόψη τις δημογραφικές αλλαγές στην αγορά εργασίας. Θεωρούμε ότι θα επέλθει βελτίωση σε αυτή την ε, νομική διαδικασία, νομοθετική διαδικασία. Μία άλλη προτεραιότητα για τα θεσμικά όργανα και τα κράτη-μέλη είναι η καλύτερη νομοθέτηση. Η Βουλγαρική Προεδρία θα ε, χρησιμοποιήσει τα δομικά υλικά που ήδη προϋπάρχουν και θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για να προσαρμόσουμε το ρυθμιστικό πλαίσιο ελέγχου και τα μη δεσμευτικά κριτήρια για την εφαρμογή των άρθρων 290 και 291 μέσα στα πλαίσια της διαδικασίας επιτροπολογίας. Τα τελευταία χρόνια τα τάχιστα βήματα στον τομέα της ε, καινοτομίας έχουν βοηθήσει την ε, ρομποτική καθώς και την ε, τεχνητή ευφυΐα που έχει μεγάλη σημασία για τη ζωή των ανθρώπων, τις επιχειρήσεις και την πολιτική. Ο, ρόλος του νομοθέτη είναι να προβεί σε μία ισβάθως ανάλυση των ε, νομικών και δεοντολογικών θεμάτων που άπτονται του τομέα της ρομποτικής και των εφιών ψηφιακών λύσεων και θα πρέπει να προωθήσουμε και τις νέες τεχνολογίες, των... Ε, 21ο αιώνα. Κατά, το άτυπο, ε, κατά την άτυπη συνεδρίαση των ε, Υπουργών Δικαιοσύνης στην ε, Σόφια, είχαμε μία πρώτη ανταλλαγή απόψεων σε ένα γεύμα εργασίας σε σχέση με την προώθηση της τεχνητής νοημοσύνης και της ρομποτικής γιατί έτσι θα είναι ευκολότερη η πρόσβαση στη δικαιοσύνη, η δικαιοσύνη θα κινείται ταχύτερα και θα λάβουμε υπόψη και τις δεοντολογικές πτυχές που συμβαδίζουν με την εφαρμογή αυτών των νέων τεχνολογιών στον τομέα της δικαιοσύνης. Κυρίες και κύριοι, Έχουμε μεγάλο φόρτο εργασίας, αντιμετωπίζουμε πολλές προκλήσεις, αλλά η ομάδα μου και εγώ, καθώς ε, και οι Υπουργοί Δικαιοσύνης, θα συνδράμουμε στη διαδικασία βελτιστοποίησης και είμαστε πεπισμένοι ότι εσείς οι Ευρωβουλευτές θα βρείτε επικοδομητικές λύσεις για όλα αυτά τα θέματα. Πιστεύω ότι θα φτάσουμε σε μία συμφωνία έτσι ώστε να προωθήσουμε τις ελευθερίες, την ασφάλεια και τη δικαιοσύνη. Ξέρετε ε, ότι το γνωμικό μας είναι ε, η εν τη ενώση. Πιστεύουμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Επιτροπή και το Συμβούλιο, όλα τα θεσμικά όργανα όταν συνεργαζόμαστε, μπορούμε να βρούμε κοινέ εξισορροπημένες λύσεις που θα ευεργετήσουν όλους τους πολίτες. Σας ευχαριστώ και θα απαντήσω σε ερωτήσεις. Ε, Ευχαριστώ πολύ για τις προτάσεις εργασίας σας, ε, κυρία Υπουργέ. Θα ήθελα να επενθυμίσω στους συναδέλφους που μόλις ε, προσήθλαν ότι μετά από την Υπουργό Δικαιοσύνης ε, της Βουλγαρίας θα δώσουμε τώρα το λόγο στον Υπουργό Πολιτισμού και μετά βεβαίως όπως κάνουμε συνήθως θα κάνουμε μια ανταλλαγή απόψεων. Έχουμε χρόνο 13 με 15 λεπτά έχετε στη διάθεσή σας κύριε Υπουργέ. Βλέπω ότι συνοδεύεστε και α, βλέπετε, μπορείτε να δείτε μάλιστα και τα ρολόγια στους ε, τοίχους. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, μέλη της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων, κυρίες και κύριοι. Είναι μεγάλη τιμή για μένα να παρίσταμε εδώ σήμερα, να παρουσιάσω τις προθέσεις μας ε, ε, στο πλαίσιο της Βουλγαλικής ε, Προεδρίας για τα θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Είναι ένα ζήτημα πολύ σημαντικό για την ανάπτυξη της καινοτομίας αλλά και της ανάπτυξης των παραγωγικών κλάδων η Βουλγαρία ανέλαβε την Προεδρία της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, σε ένα κρίσιμο σημείο. Χρειαζόμαστε περισσότερο από ποτέ ε, ενότητα, κοινέ αξίες και ένα όραμα για το μέλλον η παραγωγή και η διανομή του περιεχομένου έργων τέχνης είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο στο πλαίσιο μιας ενιαίας αγοράς και με πολύ χαρά και υπερηφάνεια θα εργαστώ επί όλων αυτών των ζητημάτων που θα έχουν αποτέλεσμα στις ψηφιακές δυνατότητες που θα προσφέρονται στους νέους ανθρώπους και σε ολόκληρη την κοινωνία. Τέσσερις τομείς προτεραιότητας. Ε, το μέλλον της Ευρώπης και οι νέοι, οικονομική ανάπτυξη και κοινωνική συνοχή, η ευρωπαϊκή προοπτική και η συνδεσιμότητα των Δυτικών Βαλκανίων, η ασφάλεια ε, και η σταθερότητα σε μια ισχυρή και ενωμένη Ευρώπη, ψηφιακή οικονομία και δεξιότητες για το μέλλον. Αυτές είναι οι προτεραιότητες μας. Η Βουλγαρική Προεδρία θα εργαστεί προς αυτή την κατεύθυνση ε, και ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να ε, συνεισφέρουμε στο όραμά μας για το μέλλον. Εμείς θα επικεντρωθούμε περισσότερο στο τελευταίο κομμάτι, την ψηφιακή οικονομία και τις δεξιότητες για το μέλλον. Θα προσπαθήσουμε να διευκολύνουμε την παραγωγή και την διανομή του ευρωπαϊκού πολιτιστικού και δημιουργικού περιεχομένου ε, με εξυγχρονισμένους και δίκαιους κανόνες για τους δημιουργούς, για τους κατόχους δικαιωμάτων και για τους παραγωγούς. Εξακολουθούμε να ασχολούμαστε με το θέμα της πνευματικής ιδιοκτησίας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό και ειδικότερα στο πλαίσιο της ψηφιακής ενιαίας αγοράς. Υπάρχει και μια πρόταση κανονισμού που αφορά για αφορά συγκεκριμένε μεταδόσεις και αναμεταδόσεις ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων μέσω ίντερνετ. Αυτό είναι ένα σημαντικό τμήμα της στρατηγικής μας τον Οκτώβριο του 2017 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τόνισε τη σημασία και την προεταιρεότητα αυτών των δύο φακέλων ε, και ότι χρειάζεται ε, περαιτέρω ε, σημαντική πρόοδος. Εμείς θέλουμε να έχουμε ένα εναρμονισμένο ευρωπαϊκό πλαίσιο στην πνευματική ιδιοκτησία που θα είναι προσαρμοσμένο στην ψηφιακή εποχή. Αυτό βέβαια έχει άμεση σχέση και με την κοινή δήλωση για τις ε, νομοθετικές προτεραιότητες των τριών θεσμικών οργάνων, Κοινοβούλιο, Συμβούλιο και Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για το 2019. Οι τρεις προηγούμενες προεδρίες ε, Σλοβακία, Μάλτα ε, και Εστονία ε, δούλεψαν πολύ σκληρά για να υπάρξει απόφαση επί των θεμάτων αυτών ε, και για ένα τμήμα που αφορούσε την πνευματική ιδιοκτησία και πράγματι προχώρησαν πολύ, γι' αυτό έχουμε μια πολύ καλή βάση για να συνεχίσουμε τη δουλειά μας για τα θέματα αυτά να επεκταθώ λιγάκι σε σχέση με αυτές τις νομοθετικέ προτάσεις και για το τι έχουμε σκοπό να κάνουμε κατά του ερχόμενου μήνες. Το Δεκέμβριο του 2017 ε, η Επιτροπή Μονίμων Αντιπροσώπων ε, συμφώνησε επί εντολή για την έναρξη διαπραγματεύσεων για τον κανονισμό ε, πνευματικών δικαιωμάτων για τις μεταδόσεις και αναμεταδόσει στο ίντερνετ ραδιοτηλεοπτικών, ραδιοτηλεοπτικού περιεχομένου και ένα από τα βασικά στοιχεία είναι η ιδέα της αρχής προέλευσης. Η θέση του Συμβουλίου είναι να συνδεθεί αυτή η αρχή με τα προγράμματα που έχουν να κάνουν ε, με ε, ειδήσει ε, και με την ραδιοτηλεοπτική μετάδοσή τους. Από την άλλη υπάρχουν οι αθλητικές εκδηλώσεις και άλλα έργα και άλλα προστατευόμενο και άλλου είδους προστατευόμενο περιεχόμενο. Τα στοιχεία ε, του νομοθετήματος αυτού ε, ενέχουν κάποια σημεία που ενδεχομένως ανησυχούν ε, τους δημιουργούς. Δεν υπάρχουν υποχρεώσεις για το διασυνοριακό επίπεδο των ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών. Μπορούν να, κάνουν, να δίνουν άδειες με όποιο τρόπο θέλουν και με γεωγραφικό αποκλεισμό. Εμείς θέλουμε να υπάρξουν τέτοιου είδους δικαιώματα ε, για όσους θέλουν να ε, μεταδώσουν μέσω ε, ίντερνετ ένα περιεχόμενο σε κάποιο άλλο κράτος μέλος. Από την αρχή λοιπόν του 2018 έχουμε κάνει τριμερείς διαλόγους. Ο πρώτος ήταν στις 20 Φεβρουαρίου. Να ευχαριστήσω τον κύριο Σφόμποντα και τους κυρώδεις εισηγητές για την επικοδομητική μας συνεργασία κατά τη συνεδρίαση αυτή. Είμαι πεπισμένος ότι η συνεργασία μας στο μέλλον θα είναι πολύ χρήσιμη και θα έχουμε έναν πολύ καλό συμβιβασμό που θα οδηγήσει σε ισορροπία μεταξύ των διαφόρων ε, ε, συμφερόντων. Να περάσω τώρα ακριβώ ε, στην πνευματική ιδιοκτησία στο πλαίσιο της ψηφιακής ενιαίας αγοράς. Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε με πολύ υπεύθυνο τρόπο, επικεντρωνόμαστε σε συζητήσεις προκειμένου να βρούμε κοινέ θέσεις, κοινό έδαφος για τα δύο βασικά ζητήματα τα οποία δεν έχουν επιληθεί, που είναι το άρθρο 11 που προβλέπει προστασία των ε, δημοσιεύσεων του τύπου σε ψηφιακές ειδήσει. Ε, προσπαθούμε να υπάρχει ένα δικαίωμα για τους εκδότες και το άρθρο 13 που θέλει να λύσει το πρόβλημα του ε, κενού αξίας δηλαδή υποχρεώσεις για τη χρήση περιεχομένου που αφορά τα το προστατευόμενο περιεχόμενο ε, λόγω της πνευματικής ιδιοκτησίας εκείνου που δημοσιεύει το περιεχόμενο αυτό. Είναι πιο αργή η πρόοδος σε αυτό το θέμα. Οι συνομοθέτες ε, δουλεύουν πολύ εντατικά. Όταν το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο θα καταλήξουν σε συμφωνία και θα έχουμε εγκρίνει τις εντολές, θα αρχίσουμε τις διοργανικές διαπραγματεύσεις και ελπίζουμε ότι αυτό θα γίνει στο δεύτερο εξάμεινο του έτους. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον Άξελ Φως για την ε, υψηλού επίπεδου δουλειά του και την ε, αφοσίωσή του στο θέμα αυτό και πιστεύω ότι θα καταλήξουμε σε κοινέ λύσεις ώστε να υπάρξει ένα νομοθετικό μέσο που θα αντανακλά τις τρέχουσες εξελίξεις και αλλαγές στο ψηφιακό περιβάλλον και που θα είναι παρκές για το μέλλον. Θα μπορεί συνεπώς να χρησιμοποιηθεί από τους δημιουργούς, τους χρήστες και τους ε, μεταδότες ε, ψηφιακού προεριεχομένου με παροχή προστασίας, ε, ισότιμης μεταχείρισης και νομικής ασφάλειας. Να σας αναφέρω τώρα και μερικά πράγματα για ένα άλλο πολύ, σημαντικό νομοθετικό ζήτημα, συνθήκη Μαρακές, που διευκολύνει την πρόσβαση στις δημοσιεύσεις για τους όσους έχουν προβλήματα όρασης, τους τυφλούς και άλλους ε, με ε, αναπηρίες. Όσον αφορά την εφαρμογή λοιπόν, ε, της της ε, συνθήκης ε, που υπεγράφει τον Οκτώβριο του 2017. Στις 17 Φεβρουαρίου εμείς αποφασίσαμε να ε, κυρώσουμε τη συνθήκη. Είμαστε τώρα στη διαδικασία της κύρωσης σε πολλές χώρες. Θα ήθελα να αναφερθώ ειδικότερα στη συνεργασία με τη δική σας Επιτροπή. Θα ήθελα να συνεργαστώ με τους εισηγητές για, τα, για τις σχετικές εκθέσεις. Είμαι πεπισμένος ότι ε, το πνεύμα συνεργασίας, ε, επικοδομητικής συζήτηση και ε, ακούγοντας ο ένας τον άλλον μπορούμε να καταλήξουμε σε πολύ θετικά αποτελέσματα. Η ποιότητα και η ταχύτητα εξέβρεσης λύσεων είναι πάρα πολύ σημαντικές και γι' αυτό θα κάνω ό,τι μπορώ για να συμμετέχω σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Υπουργέ. Επτά λεπτά. Ναι, πράγματι πρέπει να σας ανταμείψουμε γιατί πράγματι δεν ε, εξαντλήσατε το χρόνο σας. Σας ευχαριστώ που μας ε, αναπτύξατε το πρόγραμμα της Βουλγαρικής Προεδρίας. Ως ήθιστε λοιπόν τώρα οι βουλευτές, οι συναδελφοί μου, μπορούν να σας θέσουν ερωτήσεις και θα ξεκινήσουμε ευθύ αμέσως με την κυρία Κάουφμαν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να καλωσορίσω θέρμα την Υπουργό και τον Υπουργό. Καταρχάς, να πω ότι θέλω να σας ευχηθώ κάθε επιτυχία για το εξάμεινο της Προεδρίας, να σας ευχαριστήσω για τις εισαγωγικές σας παρεμβάσεις. Πράγματι, έχετε αναφερθεί σε πολύπλοκους τομείς. Ήθελα να κάνω κάποιες ερωτήσεις σε σχέση με έναν δύο τομείς. Μια πρώτη ερώτηση έχει να κάνει με την αφαιρεγγιότητα και είπατε ότι στην ομάδα εργασίας του Συμβουλίου γίνεται συζήτηση για το ζήτημα αυτό και η Προεδρία σας θέλει να επιτελεστεί πρόοδος. Θα ήθελα να μας πείτε ποια είναι τα σημαντικότερα σημεία για τα κράτη-μέλη στον τομέα του δικαίου περιφερειακότητας. Και μια δεύτερη ερώτηση. Θα με ενδιέφερε να μου πείτε κατά πόσον ε, ενδιαφέρει μόνο το πρίσμα και οπτική γωνία των επιχειρήσεων ε, αλλά και ε, των αναδιαρθρώσεων και των διαδικασιών ε, αφαιρεγκαιότητας η κήρυξη σε πτώχευση από το πρίσμα των εργαζομένων. Το δεύτερο θέμα ε, που θέλω να σχολιάσω και δεν το αναφέρατε εσείς, αλλά για μας το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο είναι πολύ σημαντικό, είναι η προστασία των καταγγελόντων. Είχαμε μάλιστα πρόσφατα ψηφίσει μια έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με πολύ μεγάλη πλειοψηφία, διότι για μας είναι πολύ σημαντικό στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να γίνει ένας κοινός προβληματισμός για να μπορέσουμε να προστατεύσουμε καλύτερα στο μέλλον τους ε, καταγγέλλοντες, τους πληροφοριοδότες. Έχουν ένα σημαντικό ρόλο στην ε, κοινωνία διότι αποκαλύπτουν, ξεσκεπάζουν ε, κάποιες παρατυπίες ή παρανομίες. Και νομίζω ότι είναι σημαντικό να ληφθεί υπόψη ο δημόσιος ρόλος τους Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω από αυτού. Υπάρχει συζήτηση στο Συμβούλιο ε, να ζητηθεί δηλαδή δράση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όπως έχουμε ζητήσει εμείς από ε, την Ευρωπαϊκή στο δηλαδή να κατατεθεί μια νομοθετική πρόταση για την προστασία των καταγγελόντων. Ποια είναι η άποψη του Συμβουλίου. Και ένα τρίτο ερώτημα, αν μου επιτρέπετε, προς τον Υπουργό Μπάνοφ μιλήσατε για, τις, ε, για τα πνευματικά δικαιώματα, ε, για τον ψηφιακό τομέα. Συνάδελφος Άξελ Φως, δυστυχώς δεν είναι σήμερα εδώ, όμως πράγματι το θέμα αυτό συζητείται εντατικότατα εδώ στο Κοινοβούλιο. Είναι ένα πολύπλοκο, δύσκολο θέμα, όλοι το γνωρίζουμε. Αναφερθήκατε στο άρθρο 11 και στο άρθρο 13. Θα ήθελα όμως να μας δώσετε κάποιες περισσότερες λεπτομέρειες. Ποια είναι τα βασικά προβλήματα που έχουν προκύψει στις συζητήσεις μεταξύ των κρατών μελών στον τομέα αυτό. Υπάρχουν εναλλακτικέ διαφορετικές για την εξέβριση πρακτικών λύσεων. Ποιες είναι οι τάσεις σε ό,τι αφορά το άρθρο 11 για τους εκδότες και την προστασία των δικαιωμάτων τους. Ευχαριστώ την κυρία Κάφμα, ο Πρόεδρος. Προτείνω, επειδή έχουμε κάποιο χρόνο στη διάθεσή μας, να απαντήσει η υπουργό ε, τώρα και στη συνέχεια και ο κύριος Τσερεμπάνοφ. Κυρία Τσάσεβα, λοιπόν, εσείς πρώτα. Благодаря, уважаема госпожо Кауфман. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την κυρία Κάουφμαν για τις ερωτήσεις. Πράγματι, μία τις προτεραιότητές μας, και πρέπει να σας πω ότι είτε εργαζόμαστε εντατικά στον τομέα αυτό, είναι η πρόταση οδηγίας για την αναδιάρθρωση. Αφαιρεγγιότητα και τη δεύτερη ευκαιρία. Σε πρώτη ανάγνωση το θέμα συστήθηκε επί Εστονικής Προεδρίας και ήταν παρόντες οι Βούλγαροι βέβαια συμμετέχοντες ε, σε αυτήν την ομάδα εργασία. Εκεί οι Εσθονοί συνάδελφοι παρουσίασαν μία πρόταση λάβουμε υπόψη μας και τις προτάσεις της Επιτροπής θεμάτων. Ο στόχος είναι η μείωση των εμποδίων για την ελεύθερη διακίνηση κεφαλαίων. Πρόκειται για εμπόδια που προκύπτουν από τις διαφορές στα νομικά συστήματα των κρατών μελών. Ταυτόχρονα όμως, οφείλουμε να εγγυηθούμε και τα δικαιώματα των εργαζομένων, των απασχολουμένων, αλλά και τα δικαιώματα όλων των επιχειρήσεων και των μικρότερων εξ αυτών. Είπατε ποια είναι τα σημαντικότερα για τα κράτη-μέλη ζητήματα. Πρέπει να σας πω ότι θα γίνουν εννέα συναντήσεις ομάδας εργασίας για το θέμα αυτό προκειμένου να συζητηθούν όλες οι πτυχές του θέματος. Και ίσως προσθεθούν και άλλα δύο, ε, άλλες δύο συναντήσεις. Υπάρχουν ε, και εισαγγελείς ε, ειδικοί στον τομέα της ε, αφεργιότητας, της πτώχευσης που θα είναι παρόντες στις εργασίες της ομάδας αυτής εργασίας. Πρέπει να σας πω ότι είναι διαφορετικές οι διαδικασίες που ισχύουν στα κράτη-μέλη. Δεν υπάρχει ομοιογένεια. Παρ' όλα αυτά θα προσπαθήσουμε να καθορίσουμε τις ε, ενδεδειγμένες απαιτήσει ό,τι αφορά την ε, αφεγγιότητα και ξεπτόχευση, αναδιάρθρωση, φροντίζοντας να προστατευτούν τα δικαιώματα όλων των πλευρών και των πιστωτών και των ε, φιλετών, αλλά βέβαια πρώτα και πάνω απ' όλα των υπαλλήλων, των εργαζομένων, διότι οι υπάλληλοι είναι αυτοί που πλήττονται πιο πολύ όταν πρόκειται για κάτι τέτοιο, όταν βρίσκεται σε δύσκολη κατάσταση ο Θέλω να σας πω ότι η προστασία των δικαιωμάτων των ε, εργαζομένων είναι για μας προτεραιότητα και φυσικά θα λάβουμε υπόψη ε, με το δέοντα τρόπο τις διαφορές ε, που, και τις ιδιαιτερότητες που αρτηρούν στα διαφορετικά νομικά συστήματα. Φαντάζομαι συμφωνείτε μαζί μου ότι πρέπει να επιδείξουμε ευελιξία στο θέμα αυτό. Αν θέλουμε να προσδιορίσουμε τις πλέον ισορροπημένες και δίκαιες λύσεις. Δυστυχώς δεν έχω αρκετό χρόνο στη διάθεσή μου για να αναπτύξω σε βάθος όλα τα άλλα ζητήματα. Όλα βέβαια αυτά ε, θα τα συζητήσουμε, όπως είναι η πρόσβαση στις διαδικασίες κήρυξη πτώχευση, ανδιάρθρωσης και δεύτερης ευκαιρίας, διορίες, και προθεσμίσει τι μεμονωμένες προσφυγές. Δύο μήνες ζητάει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τέσσερις μήνες η Κομισιόν. Και οι απόψεις των κρατών μελών διαφέρουν σε ό,τι αφορά την προθεσμία αυτή. Θα προσπαθήσουμε να καταλήξουμε σε συνένεση. Σε ό,τι δεν αφορά τις νομικές ε, συνέπειες για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, είπε και στην αρχή ότι θα προσπαθήσουμε να εγγυηθούμε στο μέγιστο δυνατό βαθμό τα δικαιώματα των επιχειρήσεων αυτών. Συνοψίζοντας λοιπόν, εργαζόμαστε με γνώμονα την προστασία όλων όσοι ενέχονται στη διαδικασία αφαιρεγγιότητας. Για το δεύτερο ερώτημα, προστασία των καταγγελόντων πληροφοριοδοτών. Είναι ένα ζήτημα ιδιαίτερος προσφυλίος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμπεριέλαβε το θέμα αυτό στο πρόγραμμα εργασίας της για το 2017 και το 2018. Είναι πολύ σημαντικό να ενθαρρύνουμε τους εργαζομένους να ενημερώσουν, να σφυρίξουν τις πληροφορίες αυτές ε, που ε, αποκαλύπτουν, που ξεσκεπάζουν ε, παρατυπίες ή παράνομες ή αθέμητες πρακτικές. Γιατί μόνο έτσι μπορούμε να αποτρέψουμε αδικήματα, ακόμα και ποινικά αδικήματα. Τη φορά αυτή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεξάγει εκτίμηση αξιολόγηση της ανάγκης να ληφθεί τομεακή ή εγκάρσια ή οριζόντια δράση στο επίπεδο αυτό. Το Συμβούλιο περιμένει την ανάλυση της Κομισιόν σε ό,τι αφορά την ανάγκη για ανάληψη δράσης για την προστασία των πληροφοριοδοτών και η Βουλγαρική Προεδρία θα είναι έτοιμη να συνεργαστεί όταν και εφόσον λάβει την ανάλυση της Κομισιόν τους καταγγέλλοντες. Ο Υπουργός Βάνο. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, κυρία Κάουφμαν. Θέλω να σας ευχαριστήσω και εγώ για την ερώτηση. Το Συμβούλιο δεν έχει μια τελική θέση ακόμη του θέματος. Αυτό που μπορώ να σας πω από αυτό το βήμα είναι ότι σε ό,τι το άρθρο 11 νομίζω ότι αρχίζει να διαφαίνεται κάποιο ενδεχόμενο συνεννόηση, συμφωνία, ελπίζω να ευοδοθεί. Δύο είναι εναλλακτικέ, όπω γνωρίζετε. Η μία εκδοχή είναι μια ε, light εκδοχή, αν θέλετε, τη πρόταση τη Κομισιόν για το δικαίωμα των εκδοτών, να είναι δικαίωμα. Και το άλλο είναι η παροχή αδειών, σε ό,τι αφορά την εφαρμογή των αδειών. Υπάρχουν κριτήρια. για να μην γίνει δεκτή μια έκδοση για το τι περιλαμβάνεται ή δεν περιλαμβάνεται σε ό,τι αφορά την 20η περίοδο προστασίας και σε ό,τι αφορά την υπόθεση του τεκμήριο του δικαιώματος των εκδοτών. Δεν μπορώ να τοποθετηθώ. Δεν και αυτός ο στόχος. Πρέπει πρώτα να ακουστούν όλα τα επιχείρηματα των κρατών μελών και εμείς έπειτα θα έχουμε το καθήκον να, να συγκεράσουμε τις διαφορετικές αυτές απόψεις. Πάντως πιστεύω ότι οδεύουμε προς εξέβρεση λύσης. Αυτή είναι η δική μου άποψη και πιστεύω ότι μετά θα αρχίσουμε να επεξεργαζόμαστε το άρθρο 13. Αλλά δεν μπορώ να σας πω ότι εδώ έχουμε επιτελέσει κάποια πρόοδο. Γιατί το σημαντικό είναι το άρθρο 11. Να βρούμε πρώτα λύση για το άρθρο 11 και αν βρούμε μία λύση εκεί και εξισορροπηθούν τα συμφέροντα, τα διαφορετικά, αυτό θα είναι πολύ θετικό γιατί πραγματικά στοχεύουμε πολύ ψηλά και αυτό είναι το σημαντικό. Και αυτό είναι το κριτήριο. Είναι ευγενής ο στόχος μας και σημαντικός. Πιστεύω λοιπόν ότι το άρθρο 11 οδεύει προς ε, επίλυση και νομίζω ότι αυτό θα βοηθήσει να πληθούν και τα προβλήματα του άρθρου 13. Σας ευχαριστώ. Πολύ σημαντική εργασία για να επιταχύνουμε. Θα ήθελα να δώσω το λόγο σε δύο μιλητές. Ο κύριος ε, Ραντεφ πρώτα και μετά ο κύριος Ζαμίχ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ε, κυρία Σάσεβα, κύριε Μπανόφ, συνάδελφοι, Καταρχήν θα ήθελα να σας καλωσορίσω στην Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και θα ήθελα να σας συγχαρώ διότι μας μιλήσατε διεξοδικά για τις προτεραιότητες της Βουλγαρικής Προεδρίας. Συμφωνώ μαζί σας ότι η Βουλγαρία έχει αναλάβει το πιδάλιο του Συμβουλίου κατά ε, τη διάρκεια μίας περίοδου που η ενότητα και η αλληλεγγύη των κρατών μελών είναι ύψης της σημασίας για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως η ενότητα των κρατών μελών θα πρέπει να βασίζεται στην εμπιστοσύνη των πολιτών και στην αμοιβαία εμπιστοσύνη όσον αφορά τα νομικά συστήματα των κρατών μελών. Σε σχέση με τις συμβάσεις για πωλήσει ψηφιακού περιεχομένου, ποιες είναι οι προθέσεις ε, της Προεδρίας για την προστασία των καταναλωτών και την εναρμόνιση. Η ερώτηση υποβλήθηκε για τους καταγγέλλοντες δημοσίου συμφέροντας, συμφέροντος, αλλά θα ήθελα να πω ότι όταν αναφέρθηκα στην έκθεση αυτής της Επιτροπής σε σχέση με τα νόμιμα μέσα για την προστασία των καταγγελόντων, είχαμε μιλήσει για οριζόντια προστασία και όχι κατακαιρματισμένη μεταξύ κρατών μελών και αυτό θα έπρεπε να γίνει μέχρι τα τέλη του 2017. Τώρα κάνουμε έκκληση προς τη Βουλγαρική Προεδρία να δώσει μια όθηση στο ζήτημα, γιατί λόγω κατακαιρματισμού δεν μπορούμε να προωθήσουμε το ζήτημα. Από πλευράς Μάλτας το θέμα ανέκυψε και όσον αφορά το κράτος ε, δικαίου στη Μάλτα και τα συμπεράσματα μίας ε, επιτροπής που επισκέφθηκε, επιτροπής ad hoc που επισκέφθηκε τη Μάλτα, διότι οι καταγγέλλοντες θα πρέπει να μπορούν να δρουν απρόσκοπτα και να την χάνουν προστασίας. Ένα άλλο ερώτημα προς τον Υπουργό Πολιτισμού σε σχέση με την οδηγία οπτικοακουστικών ε, μέσων θα πρέπει το θέμα να σας απασχολήσει άμεσα, διότι η αρχική οδηγία υπηρεσιών σε αυτό το τομέα βασίζεται στην χώρα προέλευσης και όπως είπατε ε, θα πρέπει να εξισορροπηθούν διάφορα συμφέροντα. Δεν ξέρω κατά πόσο υπάρχει ένα χρονικό πλαίσιο δράσης. Κύριε Μπανόφ, θα αρχίσουμε από εσάς, γιατί ε, ο κύριος Μπανόφ και όλα ο συνάδελφος σας απίφθηναν άμεσα τις ερωτήσεις. Και μετά η κυρία Σάτσεβα θα λάβει το λόγο. Μπορείτε να απαντήσετε με τη σειρά που θέλετε. Κύριε Ράντεφ, σας ευχαριστώ πολύ για την ερώτησή σας. Σχετίζεται με την προστασία των καταναλωτών. Αυτή είναι η πρώτη φορά που έχουμε μία προτινόμενη εναρμόνιση για την προστασία των καταναλωτών. Και αυτό στα πλαίσια της στρατηγικής για την ψηφιακή ενιαία αγορά. Υπάρχουν δύο προτινόμενες οδηγίες. Η μία για τις συμβάσεις προμηθειών ψηφιακού περιεχομένου και η δεύτερη οδηγία αφορά τις επιγραμμικές πωλήσει και άλλες μορφές τηλεπολίσεων. Η εξέταση και των δύο οδηγιών άρχισε παράλληλα, αλλά τα κράτη-μέλη αποφάσισαν ε, ότι θα πρέπει να διευρυνθεί το πεδίο εφαρμογής της ε, δεύτερης οδηγίας. Οι καταναλωτές θα πρέπει να ευεργετούνται από το ενιαίο πλαίσιο επιγραμμικών και μη πωλήσεων και αυτό έχει μεγάλη σημασία και για τους ε, προμηθευτές. Γι' αυτό δεν βρισκόμαστε στο ίδιο επίπεδο συζήτησης στις δύο οδηγίες, αλλά θα καταβληθούν προσπάθειες εναρμόνισης για ορισμένα δικαιώματα των καταναλωτών. Καταρχήν, η συμμόρφωση των συμβάσεων ε, επιγραμμικής πώλησης και επίσης αποζημιώσεις και αντισταθμίσεις όταν ε, υπάρχει ε, μία ε, λίπουσα εφαρμογή και φυσικά και ένδικα, προσφυγή σε ένδικα μέσα. Ποιο είναι το ε, επίπεδο διαπραγματεύσεων. Για την πρώτη οδηγία άρχισε ο διάλογος ε, υπό Εστονική Προεδρία. Ο τρίτος τριμερής έγινε στις ε, αρχές, στα τέλη Ιανουαρίου και στις 6 Μαρτίου προβλέπεται ο επόμενος ε, τριμερής. Για μας το Συμβούλιο αυτό αποτελεί προτεραιότητα και θα προσπαθήσουμε να φτάσουμε σε μια συμφωνία πρώτης ανάγνωσης κατά τη διάρκεια της Προεδρίας μας και ελπίζω να μας βοηθήσει σε αυτή την κατεύθυνση το ε, Κοινοβούλιο με την υποστήριξη της Επιτροπής σε σχέση με την πώληση αγαθών. Η εργασία άρχισε το Σεπτέμβριο μετά την πρόταση της Επιτροπής και θα πρέπει να εργαστούμε συζητούμε ως προς τα ευφύ αγαθά και αυτό έχει μεγάλη σημασία για εμάς. Εδώ διαφέρουν οι απόψεις των θεσμικών οργάνων. Σε σχέση με το ποια θα είναι η ρυθμιστική οδηγία αυτών των ευφυών αγαθών, αλλά εμείς θα προσπαθήσουμε να είμαστε ευέλικτοι για να ε, ταυτοποιήσουμε την καλύτερη δυνατή λύση. Αυτές οι δύο προτάσεις, όπως είπα, αποτελούν ένα μέρος της ε, στρατηγικής για την ενιαία αγορά και οι δύο προτάσεις σχετίζονται με την μέγιστη προστασία των καταναλωτών. Άρα θα προσπαθήσουμε να φτάσουμε στην ε, μεγαλύτερη δυνατή πρόοδο. Σας ευχαριστώ κύριε Σίμαρ για την ε, πρότασή σας και Ε, θα ήθελα να ε, τονίσω ότι ε, πολλοί ομότιμοι θεωρούν ότι σε αυτό το στάδιο νομοθέτησης ορίζονται δικαιώματα προσώπων, αλλά με διαφορετικούς μηχανισμούς προστασίας. Αυτό το σχετίζεται και με την προστασία των ε, καταγγελόντων. Υπάρχουν όμως αποκλίσεις. Επίσης η νομιμοποίηση εσόδων, τα χρηματοοικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θεωρώ ότι ε, οφείλω να ε, συμμεριστώ τα δικά σας συμπεράσματα, αλλά θα πρέπει να γίνει κάποιο είδος... Ε, κωδικοποίησης για να έχουμε ένα οριζόντιο νομικό πλαίσιο για γενικότερη προστασία των καταγγελόντων. Και θα ήθελα να αναφερθώ και σε ένα άλλο θέμα που έχει μεγάλη σημασία για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, για την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών και για τη δική μας Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Το προσχέδιο γνωμοδότησης ε, της Επιτροπής σας για την ελευθερία των μέσων και τον πλουραλισμό των μέσων στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, που θα πρέπει να υποβληθεί στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ σχετίστηκε με την προστασία των καταγγελόντων έτσι ώστε να μην περιορίσουμε την ελευθερία των μέσων σε επίπεδο κρατών μελών αυτό το θέμα αποτελεί προτεραιότητα, αλλά και σε επίπεδο Συμβουλίου. Επαναλαμβάνω ότι περιμένουμε τη μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τις προτάσεις της. Εμείς το Συμβούλιο θα πρέπει να δούμε τι θα προτείνει η Επιτροπή. Ε, Θεωρώ ότι η οδηγία οπτικοακουστικών μέσων έχει την ίδια σημασία με την οδηγία ως προς τη διανοητική ιδιοκτησία. Υπάρχουν ε, πολλά θέματα κλειδιά που ε, άπτονται και των δύο οδηγιών. Νομίζω ότι έχει επιτελεστεί πρόοδος, γι' αυτό μέσα στα πλαίσια της Προεδρίας μας θεωρώ ότι θα μπορέσουμε να τελειώσουμε με τους ε, τριμερείς διαλόγους και θα έχουμε μια ισχυροποιημένη θέση. Βεβαίως το θέμα της χώρας προέλευσης είναι και το θέμα κλειδί. Νομίζω ότι όλοι υποστηρίζουμε αυτή την αρχή της ε, χώρας προέλευσης που έχει μεγάλη σημασία Υπάρχουν πολλά επιμέρους ζητήματα, αλλά ελπίζω ότι θα, ότι θα ολοκληρώσουμε με τους τριμερείς διαλόγους και θα έχουμε ένα ουσιαστικό έγγραφο. Ευχαριστώ πολύ. Τρεις τελευταίες ερωτήσεις θα ακούσουμε τώρα, οι παρεμβάσεις των συναδέλφων, πριν ολοκληρώσουμε αυτήν την πρώτη ώρα εργασιών μας, Ζήφκα, Ντελβό και Ρέγνερ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο πλέον. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Υπουργό για τις συμπληρωματικές της επεξηγήσεις που αφορούν ε, τις αλλαγές, τις τροποποιήσεις, τις βελτιώσεις που έχει σκοπό να επιφέρει στη διαδικασία πτώχευσης. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και πραγματικά έχω και εγώ την τιμή να εργάζομαι επί του θέματος αυτού στην Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Θα ήθελα να επανέλθω στο Βρυξέλλες 2. Οι ε, εργασίες στο Κοινοβούλιο έχουν ολοκληρωθεί, έχει ολοκληρωθεί και ο δικός μας ρόλος, έχουμε κάνει τη δουλειά μας ως συνομοθέτης, αλλά μας ενδιαφέρει πάρα πολύ η εξέλιξη των εργασιών στο Συμβούλιο και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν κατά τη γνώμη σας είναι δυνατό να καταλήξουμε σε μία κοινή ε, θέση κατά τη διάρκεια της Φουλγαρικής Προεδρίας. Με ενδιαφέρει ιδιαίτερος ε, τα θέματα ε, για τα οποία έθεσε ερωτήματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλιο, τα παιδιά ε, και το, το μικρότερο χρονικό διάστημα ε, επιστροφής του παιδιού στο γονέα μετά την απαγωγή του. Ε, το φυσικό περιβάλλον του παιδιού επίσης. Εμείς προτείναμε σχετικά με αυτό κάποιες διατάξεις που επιτρέπουν ε, στο δικαστήριο ή στο αρμόδιο όργανο να οδηγήσει το παιδί ε, στην ε, οικογένειά του χωρίς να βλάπτεται το παιδί. Πιστεύετε ότι αυτά τα τρία σημεία που ανέφερα θα ε, προσελκύσουν την ε, ε, προσοχή του Συμβουλίου. Κυρία Ντελβό, ευχαριστώ πολύ. Κυρία Υπουργέ, πολύ χάρηκα που άκουσα ότι κατά τη διάρκεια άτυπης συνάντησης οι Υπουργοί Δικαιοσύνης συζήτησαν το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης και της ρομποτικής Οπότε θα ήθελα να μου πείτε, σημείωσα ότι μιλήσατε για τα ζητήματα ε, τα ηθικά. Δεν, έχετε σκοπό, δεν ξέρω αν έχετε σκοπό να δώσετε συνέχεια σε αυτές τις συζητήσεις. Ε, εξεπλάγει κάπως με το δεύτερο που αναφέρατε, την πρόσβαση στη δικαιοσύνη. Αναρωτιέμαι Υπάρχει βούληση μεταξύ των Υπουργών ε, Δικαιοσύνης να καταστήσουν τη δικαιοσύνη εντελώς διεφανή, κάτι το οποίο βέβαια θα με έβρισκε σύμφωνη. Αυτό που με ανησυχεί περισσότερο, κυρία Υπουργέ, είναι ότι νομίζω ότι θα ήταν σημαντικό σε επίπεδο ευρωπαϊκό να υπάρχουν αρχές ε, και, κοινή, ε, αρχές και κανόνες κοινοί, ώστε να μπορούμε να αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες, ε, να προτείνουμε νομοθεσία και να είμαστε υποχρεωμένοι σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης εκ των υστέρων να εναρμονίσουμε. Έχουμε μία ακόμη φορά τη δυνατότητα να, να προτείνουμε κοινέ αρχές. Οπότε, έχετε σκοπό να Επιμείνεται ε, στο, προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε να μπορέσουμε ε, όλοι μαζί να συζητήσουμε αυτές τις αρχές που θέλουμε να ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, ένα ακόμη ερώτημα. Χθε έγινε μία ακρόαση στην Επιτροπή μας για τα μέσα, τους μηχανισμούς συλλογικής ένδικης προστασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί υπήρχε μία έκθεση στην Επιτροπή μας ε, ε, για ε, την έκθεση για το 2016 σχετικά με το θέμα αυτό. Αυτή η σύσταση διαπιστώσαμε ότι ισχύει ακόμη, η εφαρμογή δεν είναι πολύ καλή είναι ένα ζήτημα αρκετά επίμαχο μεταξύ των κρατών μελών και των πολιτικών ομάδων. Θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω κατά πόσο η Προεδρία ε, προβλέπει τη συζήτηση του θέματος αυτού και τη συνέχιση της έκθεσης αυτής. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Κυρία Ρέγνερ. Σας ευχαριστώ. Τρεις ερωτήσεις, αλλά σύντομα. Πρώτον, δέσμη μέτρων για το εταιρικό δίκαιο, κύριε που Φυσικά και περιμένουμε την ε, Κομισιόν. Σαφέ είναι αυτό. Ωστόσο, η ερώτησή μου είναι αν έχετε ένα χρονοδιάγραμμα προβλέψει αν ε, περιλαμβάνεται δηλαδή στο καθημερινό πρόγραμμα εργασιών ε, του Συμβουλίου. Ε, τώρα, το πρόβλημα που έχει να κάνει με την παρουσία των γυναικών στα διοικητικά συμβούλια, εμείς εδώ και καιρό έχουμε λάβει τις αποφάσεις μας και πιέζουμε το ζήτημα ε, υπάρχει αυτή η εμπλοκή. Περιμένουμε όμως να λύσει το αδιέξοδο το Συμβουλίο και να μην ε, παραμένει παρατηρητής. Υπάρχουν μέτρα και αν ναι, ε, θα ήθελα αν μπορείτε να μας αναφέρετε αυτά τα μέτρα. Και το τρίτο, η εκθέσανα χώρα για τις, ε, δημοσιο... τη δημοσιοποίηση αυτών των εκθέσεων των επιχειρήσεων. Η Επιτροπή ε, η δική μας έχει να κάνει ε, με τις προϋποθέσεις διαφάνειας, υποβολής εκθέσεων αναφορών κτλ. Και στον τομέα αυτό το Συμβούλιο επίσης κολλησιεργεί εσείς τι θα κάνετε, θα εφαρμόσετε πιέσετε, ε, θα διευκολύνετε τα πράγματα στην, ε, στο Συμβούλιο υπό την ιδιότητά σας ως προέδρων, προεδρευόντων της, ε, του Συμβουλίου. Δεν βλέπω κανέναν άλλο να θέλει να πάρει το λόγο. Τόσο ή άλλως τώρα πρέπει σιγά σιγά να ολοκληρώνουμε τη συζήτησή μας. Ήταν οι τελευταίες παρεμβάσεις και ερωτήσεις. Θα ήθελα να σας ζητήσω να απαντήσετε στις ερωτήσεις που ακούσατε. Η κυρία Τσασέφα πρώτη. Ευχαριστώ. Κύριε Σβιεύκα, για την ερώτησή σας. Για τον κανονισμό Βρυξέλλες 2α, η νέα πρόταση στόχο έχει κατά κύριο λόγο την ενίσχυση των δικαιωμάτων του παιδιού και βασίζεται στην ε, Χάρτα των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και ε, στην Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Το Συμβούλιο έχει ε, είχε πολλές συναντήσεις ήδη για το θέμα αυτό και συζητήθηκε και στο άτυπο συμβούλιο στη Σόφια. Η βασική μας προτεραιότητα είναι να επιτύχουμε τη μέγιστη δυνατή πρόοδο κατά τη, βέλγη τη Βουλγαρική Προεδρία. Δέκα συνεδριάσεις έχουμε προβλέψει της ομάδας εργασίας, ενδεχομένως να προσθέσουμε και άλλες στις ήδη προγραμματισμένες. Βεβαίως υπάρχουν αρκετά ζητήματα που ε, συζητώνται και το βασικό πρόβλημα που είναι οριζόντιο είναι το συμφέρον, το καλύτερο συμφέρον του παιδιού, κάτι το οποίο βέβαια αφορά και την ενίσχυση της διαδικασίας ακρόασης των παιδιών όταν χρειάζεται κάτι τέτοιο. Ε, επίσης συζητούμε το θέμα της τοποθέτησης των παιδιών, κάτι το οποίο πρέπει να γίνει με τη συγκατάθεση ε, του ε, υποδέχοντος ε, κράτους μέλους. Γιατί αυτό θα είχε ως αποτέλεσμα την καλύτερη εξέλιξη της διαδικασίας, την ταχύτερη, εντός των ε, ε, προθεσμιών που αναφέρατε. Πρέπει να πω ότι για την ώρα υπάρχει απόκληση απόψεων σε σχέση με τις ε, ε, προθεσμίες με τα χρονικά μας όρια δεν είναι ακριβώς ίδια με αυτά που προβλέπονται στην Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών και στη Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, ε, συγγνώμη, Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ε, εμείς θέλουμε να εξασφαλίσουμε την ταχύτατη δυνατή ολοκλήρωση των διαδικασιών όταν πρέπει να γίνεται ακρόαση των παιδιών και νομίζω ακούσαμε πολλές απόψεις και δικαστών και εξέφρασαν αυτήν την άποψη. Νομίζω ότι απάντησα στο ερώτημα του κυρίου Σβιεύκα όσον αφορά την τεχνική νοημοσύνη τώρα και τη ρομποτική. Κοιτάξτε, είναι ένα ζήτημα που εμένα με ενδιαφέρει πολύ. Γι' αυτό ε, στο άτυπο συμβούλιο στην ε, Σόφια τέλη Ιανουαρίου συζητήθηκε το θέμα. Για ποιο λόγο ανέφερα την πρόσβαση στη δικαιοσύνη. Γιατί πιστεύουμε ότι η πρόοδος και η ραγδαία εξέλιξη των τεχνολογιών ε, δίνουν πολλές ευκαιρίες επιτάχυνσης ε, της δικαστικής διαδικασίας, αλλά όταν μιλάμε τώρα για την τεχνητή νοημοσύνη και τη ρομποτική, υπάρχουν και κάποια ειδικά ζητήματα που υπησέρχονται, ε, που έχουν να κάνουν με την ανταλλαγή πληροφοριών, με την προστασία προσωπικών δεδομένων. περίμενα ότι θα ήταν προβληματικό αυτό το θέμα, αλλά είναι τόσα πολλά τα προβλήματα που χρειαζόμαστε πάρα πολύ καλή συνεργασία και ελπίζω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα συνεισφέρει στην διαδικασία γιατί χρειαζόμαστε μια κοινή θέση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να καταλήξει σε κοινή θέση για τη ρομποτική και την τεχνητή νοημοσύνη δεν πρέπει να αφαιθούν τα θέματα αυτά στην αρμοδιότητα των κρατών μελών. Πολύ δουλειά λοιπόν έχουμε μπροστά μας σε σχέση με τα δύο αυτά θέματα. Ε, υπάρχουν ε, πολλά ζητήματα που θα τονίσουμε. Την προστασία των δεδομένων, τα ψηφιακά δικαιώματα, στο πλαίσιο των ε, εταιριών ε, τεχνικής νοημοσύνης και τα θεμελιώδη δικαιώματα βεβαίως, γιατί τα θεμελιώδη δικαιώματα είναι η βάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από την οπτική γωνία της δικαιοσύνης. Όλα αυτά τα θέματα επηρεάζουν τις τομεακές πολιτικές Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά ε, ως προς τη δικαιοσύνη αυτό που είναι σημαντικό ε, και που αυτό που έχει σημασία είναι πώς μπορούν οι τεχνολογίες να βοηθήσουν τη δικαιοσύνη ε, και να λάβουμε βεβαίως υπόψη ε, τα ηθικά ζητήματα. Η επόμενη ερώτηση που σημείωσα αφορά τη συλλογική ένδικη προστασία. Η Βουλγαρική Προεδρία γνωρίζει πολύ καλά τη σημασία του θέματος αυτού και της ανάγκης ανάληψης και την ανάγκη ανάληψης δράσης. Θέλουμε λοιπόν να εξασφαλίσουμε την προστασία αυτή, την συλλογική ενδική προστασία και θα προσπαθήσουμε να θέσουμε τέτοιους κανόνες ώστε να αποτρέπεται η παραβίαση δικαιωμάτων και θα θέλαμε οι διαδικασίες να είναι πιο αποτελεσματικές και πιο χρήσιμες για τους καταναλωτές. Η ανάλυση που ε, μας παρουσιάστηκε και ε, τα σχετικά πορίσματα κατέδειξαν ότι όσον αφορά τη συλλογική ενδική προστασία, το σημαντικότερο είναι να σταματήσουν οι παραβιάσεις ε, δικαιωμάτων το συντομότερο δυνατόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σκοπό έχει να προτείνει αναδιατύπωση της οδηγίας 2009 ε, κάθετος 22 και όταν ε, θα υποβληθεί η πρόταση αυτή θα αρχίσουμε να την δουλεύουμε ευθύς αμέσως. Ελπίζουμε όμως ότι αυτό θα γίνει τον Απρίλιο ότι τότε θα λάβουμε την αναθεωρημένη πρόταση και μόλις τη λάβουμε θα αρχίσουμε να την επεξεργαζόμαστε. Επίσης, περιμένουμε και την πρόταση για το εταιρικό δίκαιο και ελπίζουμε να αρχίσουμε να την εξετάζουμε το συντομότερο δυνατόν. Θα ήθελα επίσης να πω ότι πρέπει να προστατεύσουμε τα ε, δικαιώματα των εταιριών, αλλά πρέπει να γνωρίζουμε ότι και το σχετικό δίκαιο στα διάφορα κράτη-μέλη παρουσιάζει μεγάλες διαφορές. Θα προσπαθήσουμε να επικεντρωθούμε σε πολλές πτυχές όταν θα λάβουμε την πρόταση, ψηφιοποίηση για παράδειγμα, η ομάδα εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα πρότεινε την ηλεκτρονική καταγραφή, την ηλεκτρονική εγγραφή. Κάποιες χώρες όμως το φοβούνται αυτό γιατί θα καταργούσε την ανάγκη πιστοποίηση εγγράφων από τους συμβολεογράφους. Όμως αυτό είναι ένα τεχνικό ζήτημα. Και κατά τη συζήτηση της νομοθετικής πρότασης θα συζητήσουμε βεβαίως και αυτά τα θέματα. Η δεύτερη κατηγορία ζητημάτων στο πλαίσιο αυτό αφορά τις ε, διασυνοριακές ε, ε, συγχωνεύσεις Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ήθελε να ενισχύσει αυτή τη δυνατότητα διασυνοριακών συγχωνεύσεων και διασπάσεων ε, εταιριών. Ε, το θέμα, ας πούμε, της μεταφοράς της έδρας μιας εταιρείας είναι ένα σημαντικό ζήτημα. Υπό ποιες συνθήκες θα γίνεται το δικαστήριο. Έχει ε, παραγάγει μεγάλη εκτενή νομολογία ως προς αυτό και όπως έχω ήδη πει πολλές φορές, είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε, ε, να εξετάσουμε την πρόταση αυτή μόλις τη λάβουμε. Πρέπει πάντως οπωσδήποτε να εγγυηθούμε την ελευθερία μετακίνησης. Από τη μία να προστατεύσουμε τα συμφέροντα των εταιριών και από την άλλη να προσπαθήσουμε να είμαστε ευέλικτοι ως προς την εναρμόνιση των διαφόρων νομικών συστημάτων που υπάρχουν στα διάφορα κράτη-μέλη. Η ισορροπημένη εκπροσώπηση των φύλων. Αυτό είναι η επόμενη ερώτηση που έχω σημειώσει. Δύο νομοθετικές προτάσεις υπάρχουν. Ο Πρόεδρος διακόπτει λέγοντας, αν ακούμε καλά, ότι έχουμε ακόμη 15 λεπτά στη διάθεσή μας και πρέπει να ολοκληρώνουμε. Σιγά σιγά. Δύο φράσεις θα πω απλώς. Συγγνώμη που μακρηγόρησα τόσο πολύ, ε, απαντώντας τις ερωτήσεις. Δυστυχώ, αυτή η νομοθετική πρόταση που αφορά την ίση εκπροσώπηση των ε, φύλων έχει μπλοκάρει, αλλά κρατημέλη κράτη-μέλη προσφάτως ε, έδειξαν ότι μετακινούνται ως προς τις αρχικές τους ε, θέσεις και ελπίζουμε να ξαναρχίσουν οι διαπραγματεύσεις το συντομότερο δυνατόν. Πρέπει να κινητοποιήσουμε πραγματικά όλες μας τις δυνάμεις και όλους, όλους μας τους πόρους για να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μια κοινή λύση και να ε, συνεχίσουν οι διαπραγματεύσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ερωτήσεις και συγγνώμη που μακρηγόρησα. Μην ε, ζητάτε συγγνώμη. Το σημαντικό είναι να είστε συγκεκριμένοι, ακριβείς, το οποίο και πράξατε. Δώσαμε στη συζήτηση άλλα 15 λεπτά γιατί θεωρήσαμε ότι αφού είναι η πρώτη σας παρουσία στην Επιτροπή μας ε, καλό είναι να είχατε παραπάνω χρόνο. Αυτή τη φορά γι' αυτό δώσαμε ένα τέταρτο παραπάνω στη συζήτηση. Δίνω δύο λεπτά στους συναδέλφους για να βάλουν τις ηλεκτρονικές τους κάρτες ε, και θα επανακάμψουμε αφού ε, ξεπροβοδίσουμε καταρχάς ε, την Υπουργό ε, Προεδρεύουσα, την κυρία Ζιάσεφα και τον ε, κύριο Μπάνοφ Υπουργό Πολιτισμού και φαντάζομαι ότι σε αυτό το τριμηνό που απομένει θα τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ εκ μέρους της Επιτροπής. Σας εύχομαι ε, καλή τύχη και καλή επιτυχία γιατί υπάρχουν πιεστικά ζητήματα. Και τρίτον, ο πρόεδρος Βόποντα που χρειάστηκε να επανήλθει στην Πράγα και μου ζήτησε να προεδρεύσω, σας στέλνει θερμούς χαιρετισμούς. Αυτά σας χαιρετώ και σε δύο λεπτά θα ξεκινήσουμε με τις ψηφοφορίες.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 Chers collègues, je vous remercie de fermer les portes, ce qui est fait. Ε, περνάμε στις ψηφοφορίες. Ελπίζω να έχετε όλοι τις ηλεκτρονικές σας ε, κάρτες και θα υπάρξει ηλεκτρονικός έλεγχος εκεί που χρειάζεται. Αρχίσουμε λοιπόν με την έκθεση Χαουτάλα. Ψηφίζουμε την τροπολογία υπαριθμών 1. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Θέλετε να επαληθεύσουμε. Εντάξει, επαληθεύουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Λείπει μία ψήφος. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Ζητώ συγγνώμη, δεν θα προτρέξω άλλη φορά. Σας ευχαριστώ για την επαλήθευση. Συμβαστική ένα υπέρ. Κατά. Αποχές. Ε, νομίζω ότι εγκρίνεται. Τροπολογία 4. Υπέρ. Με συγχωρείτε. Α, όχι, συμβαστική 2. Με συγχωρείτε, συμβαστική 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 3. Υπέρ. Κατά αποχές ε, εγκρίνεται. Συμβαστική 4 υπέρ. αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 13. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 36. Α, όχι, όχι. Συμβαστική 5, με συγχωρείτε. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Περνάμε τώρα στην τροπολογία 38. 39, 40 και 40, ε, α, όχι, 38, 39, 40 που είναι ταυτόσιμη υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνονται. 41 υπέρ. Κατά. αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 6 υπέρ. Κατά αποχές ελέγχουμε. Φαίνεται ότι απορρίπτεται, αλλά δεν είμαι και σίγουρος. Λοιπόν, 6. Συμβαστική 6. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισατε όλοι. Ψήφισε πολύ. Πέρασε. Απορρίπτεται. Τροπολογία. Amendement numéro 22. 22. Qui est pour Υπέρ. Με συγχωρείτε, ξαναρχίζω. Υπέρ της 22. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Le 25. 25. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 35 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 43 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 45. Άμε συγχωρείτε. 47 υπέρ. Κατά αποχές φαίνεται ότι απορρίπτεται αλλά ελέγχουμε ηλεκτρονικά έρχεται η ψηφοφορία ψηφίσατε όλοι πέρας απορρίπτεται πράγματι Alors, vient maintenant l'amendement 48. 48 υπέρ. κατά αποχές εγκρίνεται 50 υπέρ κατά αποχές επαληθεύουμε άρχιδη ψηφοφορία ψηφίσατε όλοι πέρας απορρίπτεται 51 υπέρ κατά αποχές επαληθεύουμε αλλά μάλλον απορρίπτεται άρχεται η ψυχοφορία, ελέγχουμε την 51 απορρίπτεται 68 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 80. Α, όχι, καταπίπτει. 44. 44 υπέρ. Παρακαλώ να είσαστε σαφέστεροι. Είμαστε στη 44. Καταπίπτει. Γιατί? γιατί εγκρίθηκε η 13. Ωραία. 42. Καταπίπτει συμβαστική 7. Συμφωνούμε εντάξει. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 100. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 52 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 53 υπέρ κατά αποχές δεν σαφές επαληθεύουμε 53 ψηφίσατε όλοι απορρίπτεται

Φαίνεται ότι εγκρίνεται, αλλά θέλω να επαληθεύσουμε. Επαληθεύουμε την 57 άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας απορρίπτεται. 58. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 59. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 61 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Θέλετε να επαληθεύσουμε, ελέγχουμε την 61 άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι πέρας. Απορρίπτεται. 62 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν είναι σαφές. Ελέγχουμε την 62. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. 63 υπέρ. Καταπίπτει 63. 64, 65. Ωραία. Α, 60 ε, υπέρ. 66 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν είναι απόλυτα σαφές. Ελέγχουμε την 66 παρακαλώ. Ηλεκτρονικά. Tout le monde a voté, manque encore trois votes. Λοιπόν, ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Α, ε, δύο υπολείπονται. Δύο. Εντάξει, επιλογή σας. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 8 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Περνάμε στην 60 υπέρ κατά αποχές δεν είναι σαφές ε, ελέγχουμε την 60 άρχεται η ψηφοφορία Του βοτ. Ψηφίσατε όλοι. Ωραία. Πέρας. Εγκρίνεται. 67. Υπέρ. Κατά. Αποχές. ηλεκτρονικά. 67 ελέγχουμε, άρχεται. Ψηφίσατε όλοι πέρας. Απορρίπτεται. 82. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 83 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 88 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ενενήντα. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 91 υπέρ. Κατά. Α, κινήθηκα πολύ γρήγορα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν είναι σαφές. Άρχεται η ψηφοφορία για την 91. 91 ψηφίσατε, πέρας απορρίπτεται. 92 υπέρ. Κατά. Ποιοι είναι κατά. Δεν είναι σαφές. Ευχαριστώ. Αποχές. Ακόμα λιγότερο σαφές. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά για την 92. Άρχεται. έρωες, Απορρίπτεται. 95. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 96. Υπέρ. Κατά. Κατά. Κατά. Κατά. Κατά. Αποχές. γιατί το κατά είναι σαν καμπύλη αεροπλάνου. Κινείται τα χέρια από πάνω προς τα κάτω. 96. Εγκρίνεται. 97. Υπέρ. Κατά. Σας ευχαριστώ. Αποχές εγκρίνεται. 98. Α, καταπίπτει, καταπίπτει. Ωραία, ελέγχουμε ηλεκτρονικά, άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι πέρας. «21 υπέρ, κανείς κατά και δύο χέ συντριπτική πλειοψηφία. Ε, να συγχαρούμε την εισηγήτρια. κυρία Χαουτάλα θέλει το λόγο. Εντάχει, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλες τις ομάδες για τη συνεισφορά τους, γιατί δείχνει ότι μία αδύναμη σχετικά γνωμοδότηση μπορεί να γίνει πολύ συνεκτική και ελπίζω η ΛΥΜΠΕ να τη λάβει υπόψη στη δική της γνωμοδότηση. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Χαουτάλα. Μπορέσατε να πείσετε πολλούς γιατί κανένας δεν αντιτάχθηκε. Διαδικαστικό, κύριε Ζέσκα. Ευχαριστώ πρόεδρε, θα ή ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να ε, πω ότι έχω την ίδια σκέψη με την Χάουντι Χάουταλα, αλλά θα πρέπει να πούμε ότι δεν μπορούμε να δεχόμαστε να εργαζόμαστε υπό τέτοια πίεση χρόνου. Θα μπορούσαμε να είχαμε αναβάλει, να είχαμε επεκτείνει την προθεσμία, γιατί όταν υπάρχουν δύο ή περισσότερες επιτροπές που συνδράμουν, θέλουμε να ε, υπάρχει περισσότερος χρόνος για να έχει κανείς και τη μετάφραση στη γλώσσα του. Ε, την ευχαριστούμε, αλλά ελπίζω στο μέλλον να εργαστούμε διαφορετικά. Έχετε δίκιο, δεν είσαστε και ο μόνος ε, που σήμερα το πρωί εξέφρασε αυτή την άποψη. Ευχαριστούμε κύριε Ζεύσκα. Περνάμε στο... στην προφορική. Είσαστε όλοι έτοιμοι. Άρχεται η ψηφοφορία για την προφορική αυτή ερώτηση. Πρόκειται για το σημείο 21 της μερίσιας διάταξης. Δύο ακόμη παρακαλώ να ψηφίσετε ένας. Ένας, δεν έχει ψηφίσει ακόμη. Αυτός ο κάποιος δεν θέλει να ψηφίσει προφανώς. Πέρασε ψηφοφορίας. 13 υπέρ, 9 κατά. Καμία αποχή εγκρίνεται. Σας ευχαριστώ. Περνάμε στην επόμενη ψηφοφορία. Νομική βάση. Το άρθρο 22 της ημερήσιας διάταξης. Άρχεται η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Encore une voix qui manque, mais peut-être... Λείπει κάποιος εκτός αν μας εγκατέλειψε οριστικά. Πέρας ψηφοφορίας. 22 υπέρ, ομόφωνα δεκτό. Επόμενες ψηφοφορίες. Η πρώτη έκθεση της κυρίας Γκέμπχαρτ, καταρχάς. Alors, les Μου λέει η γραμματεία με πολύ λογική παρατήρηση επειδή έχουμε δύο διαδοχικές εκθέσεις της κυρίας Γκέπχαρτ. Η πρώτη είναι 2016 αυτό θα ψηφίσουμε. ...2016, κάθετος 0403. 2016 κάθετος 0403 συμφωνούμε συμφωνούμε ωραία να ξεκινήσουμε την ψηφοφορία Le premier vote va porter sur un ensemble d'amendements. Έχουμε καταρχάς ένα σύνολο τρόπο λογιών που θα ψηφίσουμε από κοινού και για να είναι ξεκάθαρο ηλεκτρονικά. Τροπολογίες 1, 2, 3 και 4. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνονται 12 υπέρ, 10 κατά. Και τώρα μπορούμε να περάσουμε στην τελική ψηφοφορία αυτής αμέσως. Άρχεται η ψηφοφορία. Είστε έτοιμοι όλοι για την τελική ψηφοφορία. Πέρασε ψηφοφορία. ψήσατε όλοι. Όχι. Ναι. Τι πρόβλημα υπάρχει. 22 ήταν οι παρόντες και 20 ψήφισαν υπέρ. Το ΕΛΚ πρέπει να σφίσει μείον, κατά δηλαδή. Συγγνώμη, λυπάμαι. Πρόεδρος, ακούστε, για να είμαστε ξεκάθαροι. Ξαναρχίζει η ψηφοφορία αν δεν υπάρχει αντίρρηση. Άρχεται η ψηφοφορία λοιπόν. 22 είναι οι ψηφίζοντες, αλλά έχουν ψηφίσει 20 μόνο. Πέρας ψηφοφορία. Ευχαριστώ. 12 υπέρ, 9 κατά, μία αποχή. Εγκρίνονται. Ευχαριστούμε κυρία ε, Γκέπχερτ. Συγχαρητήρια έκθεση σας εγκρίνεται. Και δεν σταματάμε γιατί έχουμε πάρει φόρα. Θα πάμε στη δεύτερη ψηφοφορία. Ε, Τη αγαπητή Εύελιν και εδώ η έκθεση. Τα ίδια. Θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά την τροπολογία 1, την τροπολογία 2, την τροπολογία 3 και την τροπολογία 4. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι πέρα. Εγκρίνεται 12 υπέρ, μάλλον τον μπλοκ αυτό των τροπολογιών εγκρίνεται, 12 υπέρ, 10 κατά καμία εποχή και περνάμε αυτή αμέσως στην τελική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Αν ψηφίσατε όλοι πέρα τη ψηφοφορία. 11 υπέρ αυτή τη φορά. 9 αποχές, 2, μάλλον 9 κατά, 2 αποχές, αλλά εγκρίνεται. Συγχαρητήρια κυρία Γκέπχαρτ. Εδώ λοιπόν ολοκληρώθηκε η ώρα τη ψηφοφορία από τη συνάδελφη. Σε λίγο θα περάσουμε στο τρίτο σκέλος ε, της ε, σημερινή μα συνεδρίασης. Αν σα ενδιαφέρει, όμω, παρακαλώ, Παρακαλώ, κυρίες και κύριοι, πριν περάσουν στο επόμενο, παρακαλώ, παρακαλώ, υπάρχουν επισκέπτες ε, και διάφοροι άλλοι. Παρακαλώ, ησυχία. Έχω να κάνω κάποιες ανακοινώσεις από την τελευταία συνεδρίαση των συντονιστών. 8 Μαρτίου θα χειρουργηθώ, αλλά μέχρι να γίνει αυτό παρακαλώ τη γραμματεία μας να μας ενημερώσει για τις ληφθείς αποφάσεις. Ε, σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σε συνεδρίαση της 21ης Φεβρουαρίου οι συντονιστές αποφάσισαν να ορίσουν το κύριο Λεμπρετόν ως εισηγητή ε, συντάκτη γνωμοδότησης για την έκθεση ίδιας πρωτοβουλίας ε, της ΙΝΤΑ ε, για το Harnessing Globalization Trade Aspects. Επίσης οι συντονιστές αποφάσισαν ότι δυνάμει του κανόνα 141-2 δεν θα λάβουμε δράση ε, σε ό,τι αφορά την πρόσφατη απόφαση του Ιταλικού Ανώτατου Δικαστηρίου για την ε, ανανέωση σύμβασης ενός καθηγητού ξένου στην ε, Φλωρεντία. Επίσης, σε απάντηση τη, ε, προέδρου, της επιστολής του Πρόεδρου Κάβατα για τον κύριο Κεφαλογιάννη. Να αρουμε την σας κύριο Κεφαλογιάννη. Thank you, Chair. I think... Κύριε Χάουταλο. Δεν αναφέρατε ότι αποφασίσαμε να είμαστε μια απαλλαγμένη από πλαστικά μπουκάλια και ελπίζουμε και από χαρτί επιτροπή για να προσέξουμε τον περιβαλλοντικό μας αντίκτυπο. Για να απαντήσω στο πρώτο ερώτημα. Η Γραμματεία έχει καταλάβει ότι πρέπει να προετοιμάσει και να ελέγξει την τελευταία απόφαση. Την τελική απόφαση των συντονιστών. Και θα την ανακοινώσουμε την απόφαση στο επόμενο, στην επόμενη συνεδρίαση. Δεν ήταν ο πρόεδρος έτοιμος, δεν είμαστε έτοιμοι για να ανακοινώσουμε αυτό το θέμα. Oui. Συγγνώμη, λέει κύριε Δεν είναι και ο πρόεδρος εδώ. Πρέπει να τον ρωτήσουμε όμως. Εγώ από ό,τι κατάλαβα ήταν σαφή η πλειοψηφία χθε μεταξύ των συντονιστών. Σε ό,τι αφορά την νομική υπηρεσία. για τη προϊόντα. Για να ελέγξουμε δηλαδή αν είναι εντάξει νομική βάση. Το έχουμε συζητήσει δύο φορέ. Και νομίζω ότι χθε συμφωνήσαμε. Η νομική υπηρεσία πρέπει να ε, ερωτηθεί. Και δεν το είπατε εσεί τώρα. Euh, ναι, κύριε Κάφμα. Θα σα απαντήσω, με, αλλά έχετε και δίκιο ότι ήταν και σαφές χθε. Η γραμματέα. Ναι, συμφωνήσαμε όλοι. Αυτέ είναι οι ανακοινώσει των τελικών αποφάσεων των συντονιστών. Αλλά επειδή στο συγκεκριμένο θέμα είμαστε στο προσωρινό στάδιο, θέλουμε να δούμε κατά πώς θα ασχολούμαι την νομική υπηρεσία, αλλά δεν μπορούσα να το ανακοινώσω ακόμη. Επιβεβαιώνω όμως ότι ναι, έτσι ήταν τα πράγματα χθες όπως τα είπατε. Και η λήφθη απόφαση που είπατε κι εσείς. Δεν έχω καταλάβει τίποτα. Ε, νομίζω υπάρχει μια παρανέμηση ελήφθη απόφαση ότι η νομική υπηρεσία θα πρέπει να ερωτηθεί. Το λέω και το ξαναλέω. Το καταλάβαμε έτσι έγινε, εντάξει. α, ah oui, totalement... Ναι, βεβαίω. Ναι, είναι ξεκάθαρο. Δεν υπήρχε καμιά αμφιβολία χθε. Θα ερωτηθεί η νομική υπηρεσία. Ευχαριστώ. Με ένα διάλειμμα να κάνουμε. Σας προτείνω, παρακαλώ, αγαπητοί συνάδελφοι, έχουμε ένα εργαστήριο που έπεται σχετικά με την οδηγία για το copyright και την εξόρυξη χειμών και δεδομένων συγκεκριμένα θα συζητήσουμε. 11 η ώρα ξεκινάμε ακριβώς μικρό διαλυματάκι. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να καλωσορίσω τους δύο προσκεκλημένους που θα μας παρουσιάσουν σήμερα ε, το θέμα του τελευταίου τμήματος των ε, εργασιών μας, την οδηγία για το copyright ε, και για την εξόριξη δεδομένων, ο δόκτωρ Ελεών Ωρα Ροζάτη, και καθηγητής Γκέγκερ. Μπορούν και μόνοι τους να συστηθούν οι προσκεκλημένοι μας. 15 λεπτά θα έχετε στη διάθεσή σας, έκαστος και ε, ελπίζω ότι θα τα τηρήσετε. Ε, και μετά φυσικά θα γίνει ανταλλαγή απόψεων με τους συναδέλφους ευρωβουλευτές και μετά θα ακούσουμε τα συμπερίσματά σας. Κυρία Ροσέτη, από εσάς θα ξεκινήσουμε. Έχετε το λόγο. Good morning everyone. Ε, my name is Eleonora Rosati. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελεονόρα Ροζάτη λέγομαι και θα ήθελα να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την πρόσκληση ε, προκειμένου να συμβάλλω στη συζήτηση αυτή. Είναι πραγματικά και τιμή και χαρά για μένα να συνεισφέρω κι εγώ ε, τη δική μου ε, οπτική γωνία, γιατί είναι ένα εξαιρετικό, ε, εξαιρετικά σημαντικό ζήτημα, η εξόριξη δεδομένων. Μου ζητήθηκε να διερευνήσω τις τεχνικές πτυχές για την εξόριξη δεδομένων και κειμένων και θα ήθελα να πω ευθύ εξ ότι βεβαίω οι τεχνικέ πτυχέ που θα συζητήσω μαζί σα είναι αυτέ ε, που είναι η άποψη ενός δικηγόρου που ασχολείται με την πνευματική ιδιοκτησία και ε, φυσικά θα χρειαστεί απλοποίηση και ε, να δοθεί έμφαση στις πτυχές που μπορεί να δημιουργήσουν νομικά προβλήματα. Αυτό που θα προσπαθήσω να κάνω λοιπόν είναι να σας κάνω μία επισκόπηση ε, του πώς είναι η κατάσταση στο θέμα της εξόριξης δομένων και κειμένων ε, και θα αναφερθώ και στις, στα κοινά κείμενα που υπάρχουν σχετικά θα ολοκληρώσω παρουσιάζοντας διαφορετικές ε, προσεγγίσεις για το θέμα αυτό, το οποίο, τις οποίες έχουν ακολουθήσει νομοθέτες από όλο τον κόσμο. Θα ήθελα λοιπόν σε αυτό το πλαίσιο να παρουσιάσω την αμερικανική εμπειρία, την εμπειρία του Ηνωμένου Βασιλείου, που μέχρι τώρα είναι το μοναδικό κράτος μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης, που ενέκρινε ένα κείμενο νομοθετικό που αφορά την εξαίρεση της ανάλυσης ε, κειμένων ε, και είναι κάτι το οποίο πρέπει να το λάβουμε υπόψη ε, όταν συζητούμε την ευρύτερη ε, εξαίρεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το θέμα αυτό. Θα ήθελα να ξεκινήσω λέγοντας ότι ζούμε σε μια εποχή big data, μεγάλων ε, σημαντικών δεδομένων. το, τα δεδομένα παράγονται σε τεράστιους όγκους και με μεγάλη ταχύτητα. Ε, και με πολύ μεγάλη ποικιλία βεβαίως και ε, παράλληλα με αυτό το αυξανόμενο φαινόμενο ε, της ταχύτητα της νέας παραγωγής και του όγκου των δεδομένων είναι κάτι το οποίο φυσικά πρέπει συνεχώς να το αντιμετωπίζουμε. Αυτό που είναι πραγματικά εκπληκτικό είναι ότι Γενικώ θεωρείται ότι μέχρι το 2020 το ψηφιακό ε, σύμπαν θα συμπεριλαμβάνει τόσα άστρα όσα υπάρχουν στο πραγματικό σύμπαν. Έχουμε λοιπόν αυξανόμενη διαθεσιμότητα δεδομένων που πρέπει να τύχουν επεξεργασίας γιατί η αξία τους δεν είναι η, τα ίδια τα δεδομένα αλλά στην, ε, στην εξόριξη αυτής της αξίας και ένας από τους λόγους που βλέπουμε τόσο πολύ μεγάλη αύξηση στον αριθμό των δεδομένων ε, είναι ε, το χαμηλότερο επίπεδο αποθήκευσης, οι κινητές τηλεπικοινωνίες, τα κινητά δίκτυα και φυσικά το, το ίντερνετ των πραγμάτων. Όλο αυτός ο τεράστιο όγκος δεδομένων λοιπόν ε, χρη, ε, ε, την χάνει επεξεργασία με κάποιες τεχνικές που δεν μπορεί να γίνουν βέβαια χειρονακτικά και γι' αυτό ακριβώς το έγγραφο που μια ρύθμιση της εξόριξης κειμένων και δεδομένων είναι σημαντική. Στην Ευρώπη αυτό το θέμα είναι λιγότερο ανεπτυγμένο από τις άλλα μέρη του κόσμου και αυτό το είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην αξιολόγηση αντικτύπου που συνοδεύει την πρόταση για ε, μία νέα οδηγία ε, για το copyright. Ε, αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε και με τη συμμετοχή των δικηγόρων είναι να δούμε τις νομικές ε, αμφιβολίες που υπάρχουν γύρω από την εφαρμογή αυτών των πρακτικών. Κάτι ακόμη που θα ήθελα να τονίσω εξ αρχής είναι ότι βλέπουμε οι πρακτικές αυτές ε, υπάρχουν σε μεγάλο φάσμα τομέων ε, με επιχειρηματική εστίαση, ε, δηλαδή χρησιμοποιείται η εξόριση κειμένων και δεδομένων στην υπολογιστική γλωσσολογία, στην βιομετρία, στη δασοκομεία, στην τραπεζική, στο μάρκετινγκ, στις επιχειρηματικές προβλέψεις κλπ. Επειδή λοιπόν είναι τεράστια η ποικιλία όλων αυτών των δραστηριοτήτων, είναι πάρα πολύ δύσκολο να διερευνήσει κανείς τα επιχειρηματικά μοντέλα αυτών που όντως προβαίνουν σε αυτές τις πρακτικές. Από την άποψη των, κατόχων δικαιωμάτων, δηλαδή όσων είναι κύριοι του περιεχομένου στο οποίο γίνεται η εξόριξη, είναι, είναι για αυτούς λοιπόν είναι πολύ σημαντικό να είναι γνωστές αυτές οι πρακτικές. Υπάρχουν κάποιοι που θεωρούν ότι η αδειοδότηση είναι η λύση και ότι αυτό πρέπει να γίνεται ε, σε μια καταπερίπτωση βάση και υπάρχουν κάτοχοι ε, δικαιωμάτων που επιτρέπουν την πρακτική αυτή ε, παρά την αδειοδότησή τους και υπάρχουν και κάτοχοι δικαιωμάτων οι οποίοι δεν ε, θέλουν, δεν ε, ζητούν καμία αδειοδότηση τουλάχιστον ε, για τα μη εμπορικά κείμενα και δεδομένα και επιτρέπουν την εξόριξη. Αυτό που θα ήθελα λοιπόν να συζητήσω μαζί σας τώρα είναι ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η εξόριξη κειμένων και δεδομένων. Πάμε στην επόμενη διαφάνεια. Προφανώς αυτό που προσπαθήσω να σας παρουσιάσω είναι μία απλοποίηση, μία απλουστευμένη εικόνα, γιατί υπάρχει τεράστια ποικιλία κειμένων και τεχνικών και είναι δύσκολο να υπάρχει ένα κοινό έδαφος ένας κοινό παρονομαστής. Τρία βασικά ε, βήματα υπάρχουν κατά την άποψή μου που είναι σημαντικά. Πρώτον, η εξασφάλιση της πρόσβασης ε, στο περιεχόμενο το οποίο θα υπόκειται ε, σε εξόριξη. Το δεύτερο βήμα, το οποίο δεν είναι πάντοτε απαραίτητο, αλλά σε πολλές περιπτώσεις είναι, είναι η εξόριξη και, ή και αντιγραφή του περιεχομένου, ώστε να γίνουν οι δραστηριότητες εξόριξης. Τρίτη διαφάνεια, επόμενη διαφάνεια, συγγνώμη, βλέπουμε το πρώτο βήμα που σας ανέφερα. πρέπει να αναρωτηθούν όσοι κάνουν την εξόριξη αν το περιεχόμενο είναι δωρεάν προσβάσιμο ή όχι. Αν μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτό ε, χωρίς να πληρώσουν κάτι, δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν κάποιες νομικές υποχρεώσεις που να συνδέονται με αυτό. Ε, αν πάμε πίσω στην προηγούμενη διαφάνεια, το περιεχόμενο, η πρόσβαση στο περιεχόμενο, αν είναι περιορισμένη, ε, τότε μπορεί να είναι απαραίτητο να υπάρξει μια άδεια. Αυτό μπορεί να δημιουργήσει δυσκολίες γιατί οι άδειες μπορεί να πρέπει να ε, υπογράφονται από πολλούς κατόχους δικαιωμάτων. Ε, είναι δύσκολο μερικές φορές να εντοπίσουμε καν αυτούς τους ε, κατόχους δικαιωμάτων και επειδή γνωρίζω το θέμα και πιστεύω ότι ε, αυτά τα προβλήματα όντως μπορεί να υπάρχουν και να ε, δημιουργούν προβλήματα. Βλέπουμε τάσεις ε, σε νομικό επίπεδο στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αναφέρουν ότι υπάρχει μία ανάγκη συγκατάθεσης από τους εμπλεκόμενους κατόχους δικαιωμάτων. Μπορεί να υπάρχουν λοιπόν ήδη κάποια προβλήματα από αυτό το πρώτο βήμα και ακόμη και αν υπάρξει άδεια, αυτό αφορά ένα περιορισμένο αριθμό δραστηριοτήτων και το να υπερβεί κανεί ε, τα όρια της ε, ε, άδεια μπορεί να σημαίνει ευθύνη στο πλαίσιο της άδεια αυτής. Επόμενη διαφάνεια. Υπάρχουν κάποια νομικά ζητήματα τα οποία μπορεί να προκύψουν και δεν θα τα πω με πολλές λεπτομέρειες γιατί οι ε, ε υπόλοιποι προσκεκλημένοι θα τα καλύψουν. Κατά τη γνώμη μου πρέπει να υπάρχει μία απλοποίηση, όμως μπορεί και εκεί να προκύψουν ζητήματα, κατά πόσο δηλαδή είναι τμήμα μιας βάσης δεδομένων το περιεχόμενο, γιατί στη βάση δεδομένων ε, υπάρχουν ορισμοί, ε, μπορεί να, είναι, να υπόκειται σε κόπηρα ή σε κάποιες άδειε και αυτό και μπορεί να υπάρχουν και άλλες, ε, άλλοι περιορισμοί. Και σε αυτή την περίπτωση ας πούμε η υπόθεση Ryanair και η απόφαση του δικαστηρίου για τη Ryanair είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Μπορεί να υπάρχουν ζητήματα με περιορισμούς λόγω του copyright, κάποιες, ε, κάποιοι περιορισμοί από άλλα, λόγω άλλων δικαιωμάτων ε, και αν Αν για παράδειγμα υπάρξει μία άδεια που θα εγκριθεί, ε, πρέπει να ληφθούν υπόψη και αυτά τα στοιχεία. Αν, βγούμε πέρα από την, ε, αν πάμε πέρα από την πνευματική ιδιοκτησία, υπάρχουν και άλλα νομικά ζητήματα τα οποία μπορεί να επισέρχονται, συμβατικά προβλήματα, ζητήματα προστασίας δεδομένων κλπ. Από διάφορες πηγές. Και από το GDPR. Είναι λοιπόν ένα περίπλοκο νομικό περιβάλλον που έχουμε να αντιμετωπίσουμε και πάμε στην επόμενη διαφάνεια και στο επόμενο βήμα που είναι η εξόριξη αυτή καθεαυτή. Ε, πάλι, χάρη πλούστευσης, θα προσπαθώ να σας πω ποια είναι τα κοινά βήματα στις ε, διάφορες, ε, στα διάφορα είδη εξόριξης. Υπάρχει μία φάση προεπεξεργασίας, ε, πρέπει να, γίνει, να μπει μία τάξη στο περιεχόμενο ε, των κειμένων και των δεδομένων για να μπορεί το κωδικοποιημένο μήνυμα να είναι εξορίξιμο από έναν υπολογιστή. Και αυτό μπορεί να σημαίνει ότι πρέπει να αλλάξει ο μορφότυπος, ε, να γίνει XML ένα κείμενο, να δούμε τι γίνεται με τους πίνακες, ε, με τις γραφικές παραστάσεις κλπ. Δεύτερον, η εξόριξη που είναι μια φάση που χαρακτηρίζεται από διάφορα βήματα και εκείνη. Δηλαδή μπορεί να υπάρχει tokenization, ε, δειγματοποίηση και αν δει κανείς ε, τι μπορεί να σημαίνει αυτό, ε, μπορεί αυτό να είναι πιο κατανοητό σε δυτικέ γλώσσε, αλλά να μην είναι τόσο κατανοητό σε μια γλώσσα όπω η κινέζικη, για παράδειγμα. Ε, Συνήθω υπάρχει ένα κλασικό μοντέλο που. Ε, ε που σημαίνει ότι ένα κείμενο ε, συμπεριλαμβάνει κάποιον αριθμό προτάσεων, ε, λέξεις με κενά μεταξύ τους κλπ. που είναι κάτι το σύνηθες για τις περισσότερες γλώσσες. Και επίσης πρέπει να υπάρξει μια ισοδυναμία τάξεων. Όλα αυτά είναι τμήμα ε, των δραστηριοτήτων που επιτρέπουν την προετοιμασία των κειμένων για την εξόριξη, δηλαδή να εντοπιστούν για παράδειγμα κάποιες, κάποια κάποιες συνηθισμένες, κάποια συνηθισμένη πεπατημένη για να γίνει η εξόριξη του κειμένου. Αν περάσουμε στην επόμενη διαφάνεια, βλέπουμε ότι όντως υπάρχουν νομικά ζητήματα τα οποία μπορεί να προκύψουν, να προκύψουν από ε, την δραστηριότητα αυτή. Είναι σημαντικό να δούμε και τις εμπειρίες ε, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης η προσέγγιση της, ε, των ΗΠΑ είναι αρκετά χαρακτηριστική. Στην, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στις Ηνωμένες Πολιτείες ε, πιστεύουν για παράδειγμα ότι η δημιουργία ενδιάμεσων ε, αντιγραφών ε, ενός περιεχομένου δεν στοιχειοθετούν παραβίαση των δικαιωμάτων και υπάρχει και σχετική νομολογία. Είναι ότι, ότι δηλαδή αντιγραφές δεν μπορούν να υποκαταστήσουν το αρχικό κείμενο και το σύνολο δεδομένων, αλλά επιτρέπει την πρόσβαση σε μη προστατευμένα αποσπάσματα του κειμένου που επιτρέπουν την εξόριξη του κειμένου και συνεπώς υπερβαίνουν το αρχικό περιεχόμενο. Δηλαδή δεν θα υπάρξει ανταγωνισμός μεταξύ των ειδών δραστηριοτήτων, αλλά κάποιου είδους ε, κυριάρχηση επί του προηγούμενου κειμένου. Ε, Υπάρχει λοιπόν μια εξαίρεση για την εξόριση κειμένων ε, το 2014. Ε, το Ηνωμένο Βασίλειο ε, το έκανε και αυτό. Η εξαίρεση αφορά μόνο τα εμπορικά κείμενα, αλλά οι δικαιούχοι είναι ο δικαιούχος είναι οποιοδήποτε ενδιαφέρεται να κάνει αυτή την εξόριξη. Δεν υπάρχει κανένας περιορισμός σε σχέση με τον κατάλογο των δικαιούχων. Η προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, προτάθηκε όντως από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, κάποιες επιτροπές ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχουν καταθέσει τροπολογίες για την τροποποίηση κάποιων διατάσεων. Φτάνω τώρα στην τελική μου διαφάνεια η προσωπική μου γνώμη είναι ότι προφανές ε, η εξόρυξη κειμένων και δεδομένων έχει ε, ένα πραγματικό δυναμικό στο πλαίσιο, ε, στην τρέχουσα συγκυρία που βασίζεται τόσο πολύ στα δεδομένα. Υπάρχουν προφανώς κάποια νομικά ζήτημα, ζητήματα γύρω από την εξόρυξη κειμένων και δεδομένων και θα έλεγα ότι μία υποχρεωτική εξαίρεση είναι μία ε, καλή πρωτοβουλία, όμως πιστεύω ότι δεν θα πρέπει να έχουμε μια πολύ περιοριστική εξαίρεξη που θα αποκλείει κάποιους δικαιούχους, ε, όχι μια εξαίρεση δηλαδή που δεν θα μπορούσε να επιτύχει το στόχο του να δώσει κίνητρα στην καινοτομία, καινοτομία που θα μπορούσε να προκύψει από πολλούς τομείς, ε, είτε που αφορά την έρευνα είτε που αφορά τον επιχειρηματικό τομέα. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Θερμό ευχαριστώ. Πρώτον γιατί ήσασταν ξεκάθαροι και αυτό θα μας βοηθήσει και εμείς ε, όταν χρειαστεί να αποφανθούμε και εμάς, μάλλον για όσους ήρθατε με καθυστέρηση να ακούσετε την κυρία Ροζάτη είναι καθηγήτρια σε συνδεδεμένη το Πανεπιστήμιο του Southampton για θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Θα ακούσουμε τώρα τον συνάδελφό της, τον κύριο Κριστόφ Γκεγκέρ, Διευθυντή του Κέντρου Διεθνών Σπουδών για την Πραγματική Ιδιοκτησία. Πολύ γνωστός, γνωστό μάλλον αυτό το κέντρο, στο Στρασβούργο συγκεκριμένα, στο Πανεπιστήμιο. ΣΕΙΠ είναι τα αρχικά του τμήματος αυτού. Έχετε και εσείς τον ίδιο χρόνο και σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πολύ. Χαιρόμαστε πολύ που μας προσκαλέσετε να σας παρουσιάσουμε τη μελέτη μας για την ε, εξαίρεση σε ό,τι αφορά την εξόριξη κειμένων ε, και δεδομένων. Ναι, με το κέντρο μας έχει την έδρα του στο Στρασβούργο, αλλά η δράση του είναι διεθνής. Οι συνάδελφοί μας ε, μιλούν αγγλικά, η γλώσσα εργασία τους είναι αγγλικά. Θα κάνω και εγώ την παρουσίασή μου στα αγγλικά και ζητώ συγγνώμη. Αλλά να πω ότι ε, όπως είπα βέβαια στο Στρασβούργο, άρα αν χρειάζεστε στην Ολομέλεια συμβουλευτικές υπηρεσίες, αν έχετε απορίες, είμαστε δίπλα. Και με τα χαρά να σας βοηθήσουμε σε ό,τι θέλετε. Πριν προσπαθώ να λειτουργήσω αυτό το μηχάνημα, αλλά δεν δουλεύει μπορείτε να βοηθήσετε. Ευχαριστώ. Πριν επισέλθω στα τεχνικά ζητήματα, γιατί το θέμα είναι τεχνικό ακόμη και για τους δικηγόρους, θα ήθελα να βάλω σε ένα πλαίσιο ε, το θέμα αυτό και να τονίσω τις βασικές προκλήσεις που είναι καλό να γνωρίζει κάποιος που δεν είναι ειδικό για θέματα copyright. Ποιοι είναι οι στόχοι. Στόχος είναι να δοθεί κίνητρο στην δημιουργικότητα και στην έμπνευση, αλλά και να εξασφαλίσει την ευρεία πρόσβαση ε, στους πολίτες και να βελτιώσει και την πολιτισμικότητα, την πολιτισμική ποικιλομορφία. Θέλουμε η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι χώρος καινοτομίας και δημιουργικότητας. Γι' αυτό χρειάζεται και το δίκαιο copyright. Δύο πράγματα χρειαζόμαστε. Προστασία και πρόσβαση. Αυτές είναι οι δύο του ίδιου νομίσματος και πρέπει να είναι εξασφαλισμένες και οι δύο. Για να τα πω γρήγορα και καθαρά. Στην πλευρά της προστασίας τα πάμε καλά. Έχουμε αποκλειστικά δικαιώματα που ορίζονται ευρεία ταινία στην οδηγία περί copyright και προσαρμόζονται εύκολα σε τεχνικές αλλαγές το δικαστήριο ερμηνεύει τις διατάξεις και τα πηγαίνει μέχρι τώρα πολύ καλά για να ενσωματωθεί κάθε νέα ψηφιακή χρήση. Όμως, σε ό,τι αφορά το επόμενο παρακαλώ, τους περιορισμούς δεν τα πάμε και τόσο καλά. Η οδηγία περί copyright ε, χρονολογείται από το 2001. Α, και να σας πω, το 2001 αυτή η εξόριξη κειμένων και δεδομένων ήταν επιστημονική φαντασία σχεδόν. Η οδηγία λοιπόν περί copyright από το 2001 ουσιαστικά καταρτίζει ένα κατάλογο περιορισμένων εξαιρέσεων που είναι προαιρετικές, δηλαδή τα κράτη-μέλη επιλέγουν κατά το δοκούν. Άρα εν τέλει δεν έχουμε εναρμόνιση στην πλευρά των περιορισμών και δεν έχουμε και ευελιξία περισσότερες αυτές εξαιρέσεις και περιορισμοί το 2001 έγιναν έχοντας υπόψη ότι η τεχνολογία ήταν αναλογική. Έχουν όμως οι εξαιρέσει και οι περιορισμοί σημαντικό ρόλο σε ό,τι αφορά τη διάδοση της γνώσης και στη δημιουργία ελεύθερων χώρων για την ανάπτυξη της δημιουργικότητας και ιδίως για την προώθηση της έρευνας στο ευρωπαϊκό περιβάλλον. Επίσης, στις περισσότερες περιπτώσεις συμπεριλαμβάνουν και τις θεμελιώδεις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που μας βάζουν ε, στο χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων στην κορυφή της πυραμίδας ελευθερία έκφρασης, ελευθερία πληροφόρησης, ελευθερία των τεχνών και των επιστημών. Ο νομοθέτης, εμείς δηλαδή, και δικαστές συμμετέχουμε σε αυτά. Ποια είναι η επίπτωση. Ότι χρειάζεται κατεπηγόντως μεταρρύθμιση του σκέλου ε, εξαιρέσεων και περιορισμών, ώστε να προσαρμοστεί στο ψηφιακό περιβάλλον. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπαθεί να το κάνει αυτό εδώ και πολλά χρόνια. Με μία πράσινη βίβλο καταρχά το 2008. Εγώ που είμαι ειδικό για τα θέματα copyright έχω αρχίσει να βαριέμαι. 15 χρόνια τα είδε και τα ίδια λέω. Διότι δεν έχει αλλάξει τίποτα έκτοτε. Το 2008 οι εξαιρέσει και οι περιορισμοί ήταν στο ε, παριθμόν ένα προτεραιότητα της Κομισιόν. Αλλά πολλά χρόνια χρειάστηκε να φτάσουμε εδώ. Τώρα φτάσαμε εδώ όμως. Ο στόχος της μεταρρύθμισης ε, του copyright είναι καλύτερη πρόσβαση στο ψηφιακό περιεχόμενο και ένα πιο σύγχρονο, πιο ευρωπαϊκό πλαίσιο για το copyright καθώς και διασυνοριακές επιγραμμικές δραστηριότητες για να έχουμε πραγματική ψηφιακή αγορά. Αυτές είναι προκλήσεις. Άρα μιλάμε για μια ιστορική στιγμή κατά κάποιο τρόπο. Και δεν θα πρέπει να χάσουμε αυτή την ευκαιρία. Επόμενη. Σε ό,τι αφορά την εξόρυξη κειμένων και δεδομένων, ε, έχουμε μία πήγουσα ανάγκη τα δεδομένα ε, μάλλον δεν προστατεύονται στο πλαίσιο του ε, νόμου περί copyright. Εγώ πήγαινα στις βιβλιοθήκες, ε, έκανα φωτοτυπίες και με, φωτο... και με μολύβι υπογράμμιζα τα σημεία που ήθελα, τα λίμματα που ήθελα. Αυτό ήταν τότε η εξόριξη κειμένων και δεδομένων. Αναζητούσαμε βασικές λέξεις, λέξεις κλειδιά και τώρα αυτό γίνεται με την τεχνολογία εξόρυξης κειμένων και δεδομένων πολύ πιο γρήγορα και βοηθάει να ε, αναπτυχθεί έρευνα πολύ καλύτερα. Υπάρχουν επιπτώσεις στον τομέα του copyright, αναπαραγωγή και για συναφείς γενικά δικαιώματα. Η καθηγήτρια Ροζάτη μίλησε για τις βάσεις δεδομένων. Άρα Υπάρχουν πολλές διαφορετικές ε, τεχνικές αναπαραγωγής. Επόμενο. Ποιο είναι το εφιστάμενο δίκαιο. Υπάρχει ένας κατάλογος ε, στην οδηγία για το copyright, για τα δικαιώματα δημιουργού. Και υπάρχουν εκεί σε κατάλογο οι εξαιρέσεις και οι περιορισμοί που καλύπτουν όμως ένα μικρό κομμάτι. Τα έχω συμπεριλάβει σε αυτή τη διαφάνεια που βλέπετε και τα συζητούμε και στο έγγραφό μας, μπορείτε να τα μελετήσετε με λεπτομέρειες. Καμία εξαίρεση δεν κοιτάει τη συνολικότερη εικόνα. Και το πλαίσιο δεν είναι σε καμία περίπτωση εναρμονισμένο. Υπάρχουν κάποιες χώρες που έχουν τις εξαιρέσεις, αναφέρθηκε το Ηνωμένο Βασίλειο, υπάρχουν και άλλοι όμως. Πρέπει να είμαστε τολμηροί πλέον. Αυτό είναι το μήνυμά μου ως καθηγητής νομικής. Μη διστάζετε. Προχωρήστε. Και τώρα, αν με επιτρέπετε, θα δώσω το λόγο στον συνάδελφό μου για να μιλήσει για την εφαρμογή σε εθνικό επίπεδο. Next slide, please. Επόμενη διαφάνεια, παρακαλώ. Επειδή δεν υπάρχει νομική ασφάλεια, ορισμένα κράτη-μέλη ενέκριναν εξαιρέσεις σε αυτό το τομέα. Το Ηνωμένο Βασίλειο το 2013 ήταν το πρώτο κράτος μέλος που ενέκρινε εξαίρεση για λόγους έρευνας μη, εμπορική, μη εμπορικής ε, χρήσης όταν υπάρχει νόμιμη πρόσβαση. Αυτό δεν αφορούσε τις τράπεζες δεδομένων. Το 2016 η Γαλλία ενέκρινε την εξαίρεση για ε, φορολογικές πηγές και για όχι ε, εμπορικές δραστηριότητες ως προς την ε, φορολόγηση, copyright, βάσεις δεδομένων, επικοινωνία και αποθήκευση επεξεργασμένων στοιχείων και κειμένων για να διασφαλίσουμε την ποιότητα έρευνας. Την 1η Ιανουαρίου 2017 ε, στην Εστονία έγινε ενεκρίθη μια εξαίρεση για πρόσωπα με μη εμπορικές δραστηριότητες, αλλά θα πρέπει να γνωστοποιούνται οι πηγές και η εξαίρεση ήταν δύσκολο να εγκριθεί την 1η Μαρτίου του 2018 θα ε, εγκριθούν εξαιρέσεις στην εξόριξη στοιχείων στη Γερμανία. Ε, όσον αφορά τις ε, βάσεις δεδομένων με βάση την πράξη περί copyright στη Γερμανία για μη εμπορικούς σκοπούς και στον τομέα της επικοινωνίας και αποθήκευσης ε, των δεδομένων και φυσικά για την εξασφάλιση της ποιότητας. Χωρίς να σας δώσω διεξοδικό κατάλογο, γίνονται συζητήσει σε άλλα κράτη-μέλη και το μήνυμα είναι ότι τη στιγμή που δεν το αντιμετωπίσουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο υπάρχει συνεχής κατακερματισμός στις εθνικές νομοθεσίες. Κάτι το οποίο έχει επιπτώσει στις διασυνοριακές ανταλλαγές δεδομένων. Και πολλές ε, επιδοτήσεις εξαρτώνται από την διασυνοριακή συνεργασία ε, και η ΣΕΙΠΗ είναι ένας από αυτούς τους φορείς στο Στρασβούργο. Επόμενη διαφάνεια παρακαλώ. Τώρα, ως προς τα νομικά χαρακτηριστικά αυτής της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έχει δεσμευτικό χαρακτήρα. Όλα τα κράτη-μέλη θα πρέπει να εφαρμόσουν αυτό το πλαίσιο. Δεύτερον, υπάρχει προστασία κατά της συμβατικής υπέρβασης και επίσης υπάρχουν και, ε, υπάρχει και μια εμβέλεια τεχνικής προστασίας. Ως προς την εμβέλεια και το πεδίο εφαρμογής της εξέριξης, η πρόταση επιτρέπει αναπαραγωγική διαδικασία εξόριξης ως προς τους δικαιούχους είναι τα ερευνητικά ιδρύματα τη στιγμή που πρόκειται για αποστολές ε, δημοσίου συμφέροντος. Επιτρέπεται η συνέργεια δημόσιου και ιδιωτικού τομέα μόνο σε ένα συγκεκριμένο βαθμό, μόνο σε ένα συγκεκριμένο σημείο. Ως προς τις επιπτώσεις θα πρέπει να υπάρχει εναρμόνιση έτσι ώστε όλα τα κράτη-μέλη να εγκρίνουν αυτή την εξαίρεση και να μπορούν να γίνουν διασυνοριακές εξε... εξορίξεις. Άρα θα πρέπει να ισχύει σε όλα τα κρατη ε, στη συνέχεια θα πληρώσει κάπως το κανονιστικό χάσμα όσον Φορά, δικαιοδοσίες η Ιαπωνία, Καναδά και Ισραήλ. Γιατί και εδώ ε, υπάρχουν ε, ειδικέ εξορίξεις προς άλλους ε, χρήστες. Αυτό που έχει σημασία είναι επίσης η προστασία ως προς τις ε, σημαντικές υπερβάσεις που γίνονται και για να λάβουμε υπόψη και τον ιδιωτικό τομέα. Δηλαδή, δεν θα πρέπει να επικρατήσουν ε, οι ιδιωτικοί φορείς. Επίσης, ε, δεν ε, επιτρέπει αποκλειστικά δικαιώματα σε συγκεκριμένους κατόχους όσον αφορά την διαχείριση και μεταπόληση αδειοδοσίας. Διαβάζοντας λοιπόν αυτά τα, το να αναγνώσει αυτά τα άρθρα και τους χειρισμούς θα είναι δυνατόν και στο μέλλον. Επίσης, η εξόρεξη δεν θα αλλάξει κάτι για τις δημόσιες αρχές, για τους δημοσιογράφους, για τα ερευνητικά κέντρα ή στην περίπτωση διαρροής δεδομένων, διαφθοράς και ούτω καθεξής. Ε, οι δημόσιοι φορείς δηλαδή δεν θα μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν αυτά τα δεδομένα παρά μόνο τα ερευνητικά κέντρα. Και τώρα θα δώσω το λόγο στον άλλο συνάδελφο. Και εγώ είμαι από το ΣΕΙΠΗ και θα προσπαθήσω να συνοψίσω το αχύτερο δυνατό σε σχέση με την συνολική αξιολόγηση αυτής της πρότασης. Πιστεύουμε ότι ο απολογισμός είναι θετικός σε σχέση με το TDM, με την εξόριξη δεδομένων, θα υπάρχει εναρμόνιση και νομική ασφάλεια και θα προωθήσουμε μία ψηφιακή ενιαία αγορά κάτι το οποίο είναι ύψης της σημασίας. Έτσι θα βοηθήσουμε και τις διαδικασίες καινοτομίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. <coughs> Όμως υπάρχουν, υπάρχει περιθώριο βελτίωσης γιατί θα μπορούσαμε να διευρύνουμε το πεδίο εφαρμογής της εξαίρεσης και δεν θα πρέπει να επιδοθούμε σε έναν αγώνα δρόμου, γιατί τα τελευταία δέκα χρόνια χρησιμοποιήσαμε και δημιουργήσαμε περισσότερα δεδομένα από ό,τι σε όλη την ε, ιστορία της ανθρωπότητας. Πώς μπορεί να γίνει αυτό. Γίνονται παρεμβάσεις για να ε, βελτιωθούν τα κείμενα και υπάρχει μια σειρά προτάσεων για να διορθώσουμε οριμένα τεχνικά σημεία, για να διευρύνουν αυτό το πεδίο. Αυτό που είναι πιο σημαντικό είναι το πεδίο εφαρμογής του δικαιούχου έτσι ώστε να περιοριστούν οι περιορισμοί και να υπάρχουν περισσότεροι δικαιούχοι όπως ισχύει στη Γερμανία και επίσης να επιτρέπουμε την αποθήκευση και την επικοινωνία στον τομέα των, της εξόριξης από τα ερευνητικά κέντρα. Επίσης, το δεύτερο βασικό σημείο είναι οι τρέχουσες παρεμβάσεις στα κείμενα για να μην υπάρχει τεχνολογική υπερίσχυση η οποία δεν προστατεύεται ε, από το copyright. Ε, ε, η κυρία Ροζάτη μίλησε για την απόφαση της Ryanair που κινείται προς την αντίθετη κατεύθυνση. Δεν θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει τεχνολογική υπερίσχυση. Τέλος αυτή είναι μια ευκαιρία να κάνουμε κάτι το πολύ σημαντικό, να αρχίσει μια συζήτηση για μια ανοιχτή ε, ρήτρα έτσι ώστε να βασιζόμαστε σε ε, ε, φορείς και δίκτες δίκαιης χρήσης και ρήτρες δίκαιης χρήσης κάτι το οποίο είναι ύψης τη σημασίας, έτσι ώστε το σύστημά μας να είναι πιο ευέλικτο και πιο προσαρμόσιο. Ε, μία ανοιχτή ρήτρα, μία ρήτρα ανοίγματο θα μας βοηθήσει να προβούμε σε ε, γενικότερη εξόριξη για να μπορέσουμε να εξεύρουμε και έτερους χρήσεις, δηλαδή να δούμε πώς μία λέξη έχει χρησιμοποιηθεί ιστορικά ή διαχρονικά. Αυτό αφορά και επιχειρήσεις που θα μπορούσαν να αναλάβουν αυτή την εργασία για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ευχαριστώ πολύ. Merci Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την προσπάθεια που κάνατε να είστε σύντομοι και μιλάω για τους ίδιους συναδέλφους που συνόδευσαν τον κύριο Γκάγκερ. Να δώσω το λόγο στους συναδέλφους που ζήτησαν το λόγο. Δεν ξέρω και αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να πάρει το λόγο. Πέντε λεπτά μπορώ να σας δώσω. Συγγνώμη, δεν μπορώ να σας δώσω περισσότερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ πιο σύντομα μπορώ να τα πω, δεν χρειαστώ πέντε λεπτά. Χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ σήμερα. Είναι σημαντικό τμήμα της, του, εξυγχρονισμού, του εξυγχρονισμού της πρότασης μας για το ε, copyright. Νομίζω ότι το πεδίο εφαρμογής ε, της πρότασής μας και ο στόχος ε, έχει πάρα πολύ καλά περιγραφεί από τους ε, προλαλήσαντες ε, εμπειρογνώμονες. Δεν χρειάζεται να μπω σε πολλές λεπτομέρειες. Να σας υπενθυμίσω απλώς ότι με την πρόταση αυτή της Επιτροπής εμείς θέλαμε να εξασφαλίσουμε πλήρη νομική σαφήνεια για ασφάλεια δικαίου για το θέμα της εξόρυξης δεδομένων και κειμένων γιατί θεωρήσαμε ότι σε αυτό το κομμάτι εντοπίσαμε τα περισσότερα νομικά προβλήματα κατά τη συζήτηση των τελευταίων ετών ε, και όταν, ε, όταν ε, ο στόχος μας είναι πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα κλπ. θέλουμε το νομικό πλαίσιο να είναι όσο το δυνατόν σαφέστερο. Το εξήγησαν άλλωστε και όσοι πήραν το λόγο πριν από μένα. Γι' αυτό αποφασίσαμε να προτείνουμε μία εξαίρεση ε, να μην ε, καλύπτεται από τις ε, συμβάσεις. Θελήσαμε να υπάρξουν κάποια μέτρα προστασίας των τεχνικών διαδικαστιών και να δούμε και να ξαναδούμε τις εξαιρέσεις που υπάρχουν από το 2011 οι ερευνητικοί οργανισμοί, τα ερευνητικά ε, ιδρύματα είναι πλέον αρκετά ε, οριοθετημένα ε, σε σχέση με το τι μπορούν να κάνουν στον τομέα της εξόρισης κειμένων και δεδομένων. Δεν νομίζω ότι κανένας, ούτε εσείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, διαφωνείτε με το στόχο. Βέβαια εσείς το, ε, το συζητάτε εδώ και 1,5 χρόνο. Φτάνουμε σιγά σιγά στη χρονική στιγμή κατά την οποία θα πρέπει να ληφθεί μια ε, απόφαση και στο Συμβούλιο. Ή έχουμε δει στο Συμβούλιο κάποια κείμενα κάπως πιο, πιο προχωρημένα. Ξέρω πάντως ότι και εσείς εργατικά, εντατικά εργάζεστε στο Κοινοβούλιο. Η συζήτησή μας αυτή τη στιγμή ε, συνίσταται το κατά πόσο ε, θα έπρεπε το φάσμα των δικαιούχων ε, πρέπει να επεκταθεί σε σχέση με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και νομίζω ότι υπάρχει μια σημαντική πτυχή που πρέπει να αναφέρω, εστιάζοντας περισσότερο στους κύριους φορείς της δημόσιας έρευνας, προσπαθήσαμε να εστιάσουμε παράλληλα και στον τομέα που διασπιστώσαμε τα περισσότερα προβλήματα, αναγνωρίζοντας όμως ότι καθαρά στον εμπορικό τομέα υπάρχουν ε, κάποιες άδειες ε, οι οποίες υπογράφονται τουλάχιστον σε κάποιους τομείς όπως τα χημικά, τα φαρμακευτικά προϊόντα κλπ. Νομίζω λοιπόν ότι στην προσπάθειά μας να βρούμε την τελική ισορροπία. Είναι σημαντικό όλοι οι εμπλεκόμενοι να καταλάβουν ότι υπάρχουν τομείς για τους οποίους υπάρχουν ε, λειτουργώντες ε, μηχανισμοί διαδικασιών και γι' αυτό πιστεύω, φαντάζομαι ότι και συνάδελφοί σας που θα πάρουν το λόγο μετά από μένα. Υπάρχει και μία συζήτηση που έχει αρχίσει στο Συμβούλιο σε σχέση με το ε, καθεστώς της εξόριξης ε, δεδομένων και κειμένων για περιεχόμενο που είναι ε, διαθέσιμο δωρεάν στο ίντερνετ. Προφανώς υπάρχουν κάποιες δραστηριότητες οι οποίες γίνονται αυτή τη στιγμή σε μία φαιά ζώνη, γιατί δεν ξέρουν κατά πόσο καλύπτονται από το copyright ή όχι, ε, γιατί δεν ξέρουν ακριβώς εάν καλύπτεται η βάση δεδομένων από την οδηγία copyright ή όχι. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει μία οδηγία, μία συζήτηση σχετικά με αυτό και πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας πάντοτε την τελική ισορροπία που θέλουμε να βρούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να Περάσουμε τώρα ε, στους Ευρωβουλευτές, κυρία Ρέντα και μετά η κυρία Γκέρλιγκερ και θα ήθελα να ζητήσω και από τους προσκεκλημένους μας ε, να απαντήσουν και να ε, περάσουν και στα συμπεράσματα τους σε σχέση με τη σημερινή συζήτηση. Κυρία Ρέντα, Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πολύ ενδιαφέρουσα ενημέρωση και τις ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις. Είναι μια ερώτηση και προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σε εσά ως ερευνητές, γιατί αναφέρατε τους δημοσιογράφους και τη χρήση της εξόριξης στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Συμφωνούμε ότι οι δημοσιογράφοι και οι εφημερίδες είναι ιδιωτικέ εταιρείε, ε, δεν είναι ερευνητικά ιδρύματα και όμως κάνουν εξόριξη δεδομένων. Σήμερα το πρωί μια μια συζήτηση με ε, έναν εκπρόσωπο στην ε, ομάδα υψηλού επίπεδου για ε, τα, τις ψευδείς ειδήσει και προσπαθήσαμε να δούμε πώς θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε την εξόριση δεδομένων για τις ψευδείς ειδήσει ε, είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό ότι κάποιος ε, δημοσιογράφος που κάνει εξόριξη θα πρέπει και εκείνος να λάβει μία άδεια για την εξόριξη ε, άρθρων ειδησεογραφικών. Επειδή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είπε ότι υπάρχουν κάποιες λύσεις αδειοδότησης για τους εμπόρους, από ποιον πρέπει να λάβουν άδεια οι έμποροι ε, συγγνώμη, οι, δημοσιογράφοι για ε, να μπορέσουν να κάνουν εξόριξη δεδομένων σε σχέση με τις ψευδείς ειδήσει, γιατί υπάρχουν ε, οργανισμοί νόμιμοι οι οποίοι προβαίνουν σε ψευδείς ειδήσει και δεν μπορώ να καταλάβω πώς ένας δημοσιογράφος θα μπορούσε να πάρει μία άδεια για να μπορέσει να ε, παροπλήσει ας πούμε ένα site, έναν ιστότοπο από ψευδείς ειδήσει. Η κυρία Γκέρλιγκερ, και εγώ θα ήθελα να κάνω μία ερώτηση. Σας δίνω και δύο λεπτάκια για να βάλετε τα ακουστικά. Πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση. Δεν είναι εδώ η συγητής όμως που ασχολήθηκε με το θέμα αυτό αλλά είμαι σκιώδης εισηγήτρια εγώ και έχουμε κάνει πολλές συναντήσεις ε, μεταξύ σκιωδών εισηγητών. Αυτό που είπατε για τις εξαιρέσεις ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Το είπατε κι εσείς και όποτε κι εμείς μιλάμε για εναρμόνιση αυτών των εξαιρέσεων. Είναι σαν να ανοίγουμε το κουτί της Πανδώρας για πολλούς. Δεν ξέρω κατά πόσον λοιπόν ε, είναι ε, και ρεαλιστικό να συνεχίσουμε να το ζητάμε αυτό. Δεν ξέρω κατά πόσον θα πραγματοποιηθεί. Ήμουν και η εισηγήτρια για το ορφανά έργα και όταν ξεκινήσαμε τις εργασίες ε, τα ίδια μας λέγανε. Μην το ακουμπάτε το θέμα αυτό, δεν πρόκειται να υπάρξει εναρμόνιση. Τελικά υπήρξε Δείχθηκε ότι ήταν δυνατόν να υπάρξει εναρμόνιση αν ο δημιουργός εμφανιστεί ανταμείβεται αλλά βρήκαμε και άλλες λύσεις άρα νομίζω ότι μπορούμε να αντλήσουμε διδάγματα από την εμπειρία αυτή και λυπούμε που δεν είναι εδώ οι πιο συντηρητικοί συνάδελφοι μεταξύ των μελών της Επιτροπής μας, δεν βρήκαν χρόνο για να έρθουν εδώ. ρωτώ όμως, επειδή το δικό σας το επάγγελμα. Ως επαγγελματίε, λοιπόν, πείτε μου. Μπορούμε να μιλήσουμε για αντίγραφα, μπορούμε να μιλήσουμε για sharing. Δεν είναι το ίδιο πράγμα ένα αντίγραφο ή αντιγραφή με αυτό που ήταν πριν 50 χρόνια. Άρα και το λεγόμενο sharing ε, δεν είναι ό,τι ήταν πριν από πολλά χρόνια. Μιλάμε για πράγματα και δικαιώματα ε, που αφορούσαν άλλη πραγματικότητα πριν από 40, 50, 60, μην και το 19ο αιώνα. Άρα τώρα χρειαζόμαστε μια εντελώ διαφορετική προσέγγιση. Δεν μπορούμε να καθόμαστε στο γραφείο μας όπως κάναμε και αντιγράφουμε ένα απόσπασμα του βιβλίου που μας ε, έδωσε η φίλη μας να διαβάσουμε. Έτσι το βλέπετε και έτσι συζητείτε με αυτό το πνεύμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπορείτε να απαντήσετε, ο κύριος Γκάιγερ, η κυρία Ρωσάτη. Εκτό εάν εκχωρήσει τι εξουσίες της σε κάποιον, σε κάποιον άλλον ο κύριο ε, Γκάγκερ. Κυρία Ρωσάτη. Συμφωνώ απολύτω με αυτό που είπατε και θα ήθελα να απαντήσω και στο σχόλιο της κυρία Ρέντα. Πράγματι, ο σημερινός κόσμος είναι πολύ διαφορετικός από αυτόν ε, που είχαμε πριν από 20 αλλά και πριν από 5 χρόνια. Υπάρχει λοιπόν μία εκθετική ε, ανάπτυξη σε πολλούς τομείς και δεν νομίζω ότι κάθε φορά η ερμηνεία του copyright ήταν πάντοτε συμβατή με αυτές τις αλλαγές που διαπιστώνουμε. Για την αντιγραφή, για παράδειγμα, αν η εξαίρεση για τις προσωρινές αντιγραφές, ε, απλώς και μόνος για να σας δώσω ένα παράδειγμα, αν ισχύει λοιπόν αυτή η εξαίρεση ε, για τα προσωρινά αντίγραφα, η ιδέα της αντιγραφής ε, νοείται ως ευρύτερη. Γίνεται μια ευρεία ερμηνεία του τι θα πει αναπαραγωγή ακόμη και αν ένα μικρό τμήμα αναπαράγεται, αυτό μπορεί να, να θεωρηθεί αντικείμενο παράβαση. Συμφωνώ με αυτό και σε σχέση με το σχόλιο της ε, κυρίας Ρέντα. Πράγματι μπορεί να υπάρχει μια κατάσταση κατά την οποία αυτοί που κυκλοφορούν σε ειδήσει να προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Μπορεί να υπάρχει λοιπόν μια κατάσταση εντελώς ε, αντιφατική. Η ιδέα το να έχουμε λοιπόν έναν πολύ στενό, πολύ μικρό και διεξοδικό κατάλογο δικαιούχων, αυτό το σκοπό εξυπηρετεί, αυτό προσπαθεί να καλύψει. Αν δεν κάνω λάθος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τόνισε ότι το κείμενο για την εξόριξη δεδομένων θεωρείται ένα εργαλείο στον τομέα της έρευνας, για παράδειγμα. Ε, επειδή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για παράδειγμα στον επιχειρηματικό τομέα και αναφέρομαι βέβαια και στη δημοσιογραφία. Αν λοιπόν κάτι έχει ήδη δρομολογηθεί, για ποιο λόγο πρέπει να περιοριστεί. Και ολοκληρώνοντας, νομίζω ότι η αναφορά στην εμπειρία του Ηνωμένου Βασιλείου και τη... νομίζω ότι είναι χρήσιμη, γιατί σε κάποια φάση τη συζήτηση στο Ηνωμένο Βασίλειο υπήρχε το ζήτημα του ποιος θα, ποιο, ποιοι θα είναι οι δικαιούχοι της εξαίρεσης. Ε, η κυβέρνηση έλαβε γνώση του ότι υπάρχει ε, μία ε, αγορά την οποία θα αφορά το θέμα αυτό αλλά κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ακόμη και αν υπάρχουν άδειες σε μερικές περιπτώσεις είναι πάρα τόσο δύσκολο να υπάρξει άδεια η έγκριση πρέπει να είναι αποτέλεσμα ε, συγκατάθεσης τόσο πολλών ε, ε, κατόχων δικαιωμάτων που αυτό θα μπορούσε να είναι ένα τεράστιο εμπόδιο που δεν μπορούμε να υπερβούμε που τελικά μπορεί να οδηγήσει στην παρεμπόδιση μιας σημαντικής έρευνας. Λοιπόν, αυτό σας το λέω γιατί πιστεύω ότι μπορεί αυτή η εμπειρία να είναι χρήσιμη και για σας. Γι' αυτό σας την ανέφερα. Είναι μια συζήτηση που δεν έγινε πριν από μεγάλο χρονικό διάστημα. Το 2014 εισήχθη αυτή η εξαίρεση. Ε, Ενδεχομένω λοιπόν να είναι πράγματι συγκρίσιμο το περιβάλλον το, ε, το τεινό με το τωρινό. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε, Σας ευχαριστούμε κύριος Γκάικερ. Δύο πολύ σύντομα σχόλια. Στο δικό μας έγγραφο δεν έχει διανεμηθεί, αλλά υπάρχουν αντίτυπα. Τόσο πάνω μπορεί να, μπορούμε να σας στείλουμε ένα ε, ηλεκτρονικά. Μπορεί να υπάρξει επέκταση του φάσματος των δικαιούχων. Αλλά δεν μας ικανοποιεί και πολύ η λογική, εκτός από ερευνητικά ιδρύματα, το σχέδιο διοδοτήσεων λειτουργεί. Έγινε κάποια αξιολόγηση, διαρωτώ. Είπε και η καθήτρια Ροζάτη ότι η εξόριξη κειμένων και δεδομένων έχει να κάνει με άδεια για τους ε, ανθρώπους που χρησιμοποιούν τα δεδομένα, που χρησιμοποιούν τα συγγενικά δικαιώματα, υπάρχει το δικαίωμα στην ιδιωτική σφαίρα κτλ. κτλ. Άρα το σχήμα αυτό, το πρόγραμμα διοδότης καθίσταται άκρος πολύπλοκο. Σήμερα λοιπόν αυτό που πρέπει να αποφύγουμε είναι να δημιουργηθεί μια εξαίρεση που καθίσταται αμέσως παροχημένη. Και για την αναθεώρηση μιας οδείας ξέρετε πόσος χρόνος απαιτείται. Αλλά εμείς θέλουμε να ανθεί η δημιουργικότητα στην Ευρώπη. Και όχι μετά από δύο χρόνια να δούμε με θλίψη ότι έχουμε μπει σε ένα κλειό που μας περιορίζει. Για κάποιες λοιπόν εμπορικές χρήσεις, για κάποιους εμπορικούς χρήστες υπάρχει πάντα μηχανισμός που γνωρίζουμε για την αμοιβή. Ίσως αυτό είναι μια συμβιβαστική λύση να ανοίξω κατάλογο των δικαιούχων. Παραδείγματο χάρη για τα press reviews. Αν επιτρέψουμε στις επιχειρήσεις να κάνουν ηλεκτρονικά αυτή την επισκόπηση για τις επιχειρήσεις μπορεί να ε, υπάρξει, να γεννηθεί δικαίωμα ε, αμοιβή. Σε ό,τι διαφορά αφορά το γεγονό ότι το αντίγραφο σήμερα δεν έχει καμία σχέση με το αντίγραφο πριν από πολλά χρόνια, ισχύει. Σήμερα κάνουν πολλά αντίγραφα. Και δεν ξέρουμε καν ότι είναι αντίγραφα. Όταν ε, σερφάρουμε στο διαδίκτυο υπάρχουν αντίγραφα που διατηρούνται στον υπολογιστή μας. Και αυτό δεν έχει να κάνει φυσικά σε καμία περίπτωση με την εκτύπωση ή την φωτοτυπία που κάνουμε ε, από ένα άρθρο μιας εφημερίδας στο φωτοτυπικό μηχάνημα. Κάποια από αυτά εντάσσονται στις αναπαραγωγές δυνάμει του άρθρου περί copyright. Όλα αυτά τα αντίγραφα που κυκλοφορούν εκεί πέρα πρέπει να βεβαιωθούμε ότι δεν δημιουργούν πρόβλημα, δεν μπλοκάρουν κάποιον ή κάτι. Δεν βλέπω να θέλει κάποιο άλλο συνάδελφό μου το λόγο. Για μια ακόμη φορά, λοιπόν, εκ μέρου Επιτροπή μα θέλω να σα ευχαριστήσω. Α, εσεί, παρακαλώ. Επειδή έχουμε λίγο χρόνο, Έχω δύο ερωτήσεις. Ίσως υπάρχει μία διάκριση μεταξύ εμπορικής και μη χρήσης, όπου η εμπορική χρήση προβλέπει και μία αντιστάθμιση για να μιλήσω για το δημοσιογράφο που προσπαθεί να αναλύσει ψευδείς ειδήσει είναι εμπορικός φορέας, μετά θα πρέπει να καταβάλει ε, ένα αντίτιμο σε αυτό που χρησιμοποίησε ή που δημιούργησε τα fake news. Αυτό μου φαίνεται πολύ άδικο θα πρέπει να προβλέπετε αποζημίωση σε περιπτώσεις όπου έχουμε να κάνουμε με επαγγελματικές ε, προσφορές. Αλλά σε αυτή την περίπτωση δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Υπάρχουν επιχειρήσεις, όπως ελέγχθη αυτή την εβδομάδα σε ένα πρόγευμα, που θέλουν να δημιουργήσουν έναν αλγόριθμο για να μπορέσει να ανοιχνεύσει ένα συγκεκριμένο παπούτσι και ε, αυτός ο αλγόριθμος ειχνηλατεί όλα αυτά τα παπούτσια στο διαδίκτυο. Αυτοί που έβγαλαν την αρχική ε, φωτογραφία δεν είναι επαγγελματίε. Εάν λοιπόν προσπαθεί κανείς να χορηγήσει αυτή την αντιστάθμιση δεν θα πρέπει να υποστεί έναν υπερβολικό διοικητικό φόρτο. Και το δεύτερο ερώτημα αφορά κάτι που συζητήθηκε στο Συμβούλιο. Μετά την εξόριξη τα αντίγραφα πρέπει να διαγραφούν. Αναρωτιέμαι ε, από πρακτικής πλευράς τι σημαίνει για την ε, αναπαραγωγιμότητα των εγγράφων και εντάσσεται στο copyright ή όχι γιατί μέσα στα πλαίσια του copyright επιτρέπεται ή δεν επιτρέπεται κάτι σαφώς δηλαδή η ε, αναπαραγωγή και η αντιγραφή, γιατί επιτρέπεται η αναπαραγωγή, αλλά για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, εκτός από την εξαίρεση γιατί η αντιγραφή επιτρέπεται σε μεταβατικά συστήματα. Δεν ξέρω λοιπόν κατά πόσο αυτή η διαγραφή έχει νόημα. πολύ ε, σύντομα παρακαλώ. Οι απαντήσεις, ε, ναι, εντάχει, ως προς το πρώτο ερώτημα, αναφέρθηκα στη δυνατότητα ανταμοιβή στα πλαίσια διεύρυνσης του πεδίου εφαρμογής. Αυτό δεν σημαίνει ότι μιλώ για δημοσιογράφους. Ας πούμε ότι έχουμε νέα startups, δηλαδή χρηματιστές που θέλουν να εξορίξουν στοιχεία για επιχειρήσεις ως προς ε, στοιχεία με εμπορική αξία για εμπορικούς σκοπούς. Αυτό είχα κατά νου τις νεόκοπες δηλαδή επιχειρήσεις. Δεν ε, μιλούσα για δημοσιογράφους. οποιαδήποτε αποζημίωση θα πρέπει να ακολουθήσει μία διαδικασία δοκιμών. Θα πρέπει να δούμε κατά πόσο πλήττεται ο ενδιαφερόμενος, για παράδειγμα. Ένα άλλο σημαντικό σημείο ως προς την αναπαραγωγή ε, να θυμόμαστε ότι όλες οι τεχνικές εξόριξεις δεν σημαίνουν και αναπαραγωγή, γιατί υπάρχει και η τακτική crawling, η οποία ε, χρησιμοποιείται ευρέως. Δεν υπάρχει διασάφηση, γιατί θεωρούμε ότι το πεδίο εφαρμογής μπορεί να είναι διαφορετικό και πρέπει να προσαρμοστούμε. If I can, uh, know, um, uh, uh, επ' αυτού θα ήθελα να προσθέσω ότι σε αυτή την περίπτωση χρειάζεται αντιστάθμιση ή αποζημίωση. Αν μιλήσουμε για το ιδιωτικό τομέα, την ιδιωτική ε, αναπαραγωγή, αυτή συνδέεται με την ίδια την ε, πράξη. Στην περίπτωση της εξόριξης τι γίνεται με το copyright. Γιατί η εξόριξη είναι κάτι που δεν θέλει να οδηγήσει σε ανταγωνισμό ή υποκατάσταση στην αγορά. Πρόκειται για, μια, ε, για ένα υπερισχύον περιεχόμενο που λαμβάνει υπόψη πτυχές που δεν προστατεύονται από το copyright, όπως ιδέες ή γεγονότα, και να τα χρησιμοποιήσουμε για να προωθήσουμε τη γνώση σε ορισμένους τομείς. Δεν νομίζω λοιπόν ότι χρειάζεται αποζημίωση. Ως προς τη διάκριση εμπορικής ημιχρήσης, αυτό ε, δεν είναι απλό και ευδιάκριτο. Και εδώ θα αναφερθώ σε έναν άλλο τομέα copyright, δηλαδή το δικαίωμα επικοινωνίας με το κοινό. Αν δούμε πώς το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ε, προέβη σε αυτή τη διασύνδεση, φαίνεται ότι μετά την απόφαση για το GS Media έχει μεγάλη σημασία να δούμε κατά πόσο ο σύνδεσμος λειτουργεί με σκοπό το κέρδος αλλά δεν ξέρουμε τι εννοούμε με το κέρδος, δηλαδή ποιος είναι ε, ο υπεύθυνος, ο link provider στην συγκεκριμένη περίπτωση. Άρα δεν είναι ευδιάκριτη η εμπορική μη χρήση στην εξόριξη. Θα πρέπει να είμαστε πολύ σαφείς και για το πότε ισχύει το ένα σενάριο ή το άλλο. Και ως προς το δεύτερο σημείο, για την πρόληψη της αποθήκευσης αντιγράφων, ξέρω, καταλαβαίνω τη λογική σας, να μην υπάρξει δηλαδή η ε, μεταγενέστερη χρήση του περιεχομένου πέρα από την εξόριξη. Δεν προβλέπεται η αποθήκευση, αλλά η νέα χρήση για στόχους πέρα της εξόρυξης. Είναι λίγο διαφορετικό λοιπόν αυτό το σημείο, το οποίο θα μπορούσε να αποσαφινιστεί αν επικρατήσει αυτή η λογική. Χρειάζεται λοιπόν σαφήνεια επί του σημείου. Έχουμε μία λύση που ισχύει στην περίπτωση της Γερμανίας, γιατί εδώ το θέμα είναι η επαλήθευση του αποτελέσματος. Μπορούμε να αποθηκεύσουμε τα αποτελέσματα της εξόρυξης σε έναν ε, ασφαλή εξυπηρετητή έτσι ώστε οποιοδήποτε ακαδημαϊκός να μπορεί να προστρέξει και να επαληθεύσει το αποτέλεσμα μέσα στα πλαίσια της επικοινωνίας και με το κοινό αλλά η αποθήκευση μπορεί να γίνει σε έναν ασφαλή τόπο. Εξ ονόματος όλων των συναδέλφων και των παρόντων θα ήθελα να ευχαριστώ τους εμπειρογνώμονες και τους πάνελιστ που σήμερα μας ε, ε, έκαναν εισηγήσεις για την εργασία τους επειδή δεν υπάρχουν άλλα θέματα στην ημερήσια διάταξη. Σας ευχαριστώ πολύ. Λύεται η συνεδρίαση της Επιτροπής μας. Καλή σας όρεξη.